Καλημέρα σας. Είχα πει ότι θα θέλω να ξεκινήσω στην ώρα μου. Ξεκινούμε λοιπόν αμέσως με το σημείο 6 της σημερισίας διάταξης. Πρόκειται για ψηφοφορία και ελπίζω να έχετε όλοι φροντίσει να φέρετε την κάρτα για την ψηφοφορία. Τοποθετήστε λοιπόν τις κάρτες σας στα μηχανήματα. Να είμαστε έτοιμοι και να ξεκινήσουμε. Έχουμε την έκθεση για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Και ξεκινούμε αμέσως με τη συμβιβαστική τροπολογία 1. C1, δηλαδή C1. Υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία, συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Συμβαστική υπαριθμών 2, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές. Εγκρίνεται σε 3. Υπέρ κατά αποχές έτσι λοιπόν έχουμε εγκρίνει τις τρεις τροπολογίες και προτείνω να περάσουμε στην, αριθμόν, στην υπαριθμόν 5, υπαριθμόν 5 τροπολογία υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 τώρα. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45. Υπέρ της 45 παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 7. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50. Υπαριθμών 50. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και περνάμε στην 54. Υπέρ της 54 παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πενήντα Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μάλλον και περνούμε στην 61, 61 τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται η 61. Και ε, γυρνάμε σελίδα για να περάσουμε στην 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εβδομήντα πέντε τώρα υπέρ κατά αποχές. Παρακαλώ. Αποχές. Εγκρίνεται. Κύριε Πρόεδρε, μια πρόταση παρακαλώ από την 75 μέχρι την 91 να ψηφίσουμε on block τις τροπολογίες ομού. Έχει τα παραρτήματα τουλάχιστον. Προτείνω λοιπόν, προτείνω από την 116 μέχρι την 144 ομού παρακαλώ τουλάχιστον. 116 με 144 να ψηφίσουμε ομού όλες τις άλλες χωριστά γιατί ε, είναι προς διαφορετικές πλευρές της ψηφοφορία καθόλου. Also was wir machen können, Frau Kollegin, ist 76 bis 81, weil 75 76 μέχρι 81 λέτε, την 76, 75 την έχουμε ψηφίσει, 76 μέχρι και 81 ομού μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ παρακαλώ, 76 με 81 κατά αποχές εγκρίνεται, ε, απορρίπτεται συγγνώμη. Στη συνέχεια έχουμε διαφορετικέ προτάσεις στι ε, στις τροπολογίε τροπολογίες, τις ψηφίσουμε χωριστά. 82 παρακαλώ υπέρ, κατά άποχες. Απορρίπτεται. 83. Υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται 84 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93 τώρα με μια διόρθωση θα την ψηφίσουμε. Την έχετε στα εγγραφά σας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ενενήντα έξι τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φτέρμα στην 100 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εκατόν 104 υπέρ κατά άποχες Εκατόν πέντε τώρα παρακαλώ υπέρ Εκατόν έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές αφορύπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 110 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 23 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίψετε Ψηφίζουμε τώρα την 111 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Περ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ για μια φορά. Υπέρ. Με τα χέρια λέει ο πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις πληροφορίες. 22 υπέρ. 31 κατά. Καμία αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα και πάμε στο 24 τώρα υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την 25 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26, παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 τώρα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 27 κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα έχουμε μια πρόταση από την 116 μέχρι την 144 να ψηφίσουμε ομού τις τροπολογίες. Έκανε πολύ σκληρή δουλειά και καλή πρόταση πολύ. Παρακαλώ να μου πείτε ποιος συμφωνεί με τις ε, τροπολογίες αυτές υπέρ κατά αποχές. Από την 116 έως και την 144 απορρίπτονται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Είναι πρώτος του εισηγητού. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 προφορική τροπολογία, με προφορική τροπολογία με την προφορική της τροπολογία λοιπόν την ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται με την, με την προφορική τροπολογία. Στην 41 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά οι σοσιαλδημοκράτες έχουν μία ψήφο περισεβούμενη. Καλώς. Κλείνει λοιπόν η ψηφοφορία. Εψήφισαν 65 υπέρ, 5 αποχές και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η επόμενη ψηφοφορία είναι έκθεση της κυρίας Χάουκ. kommen, jetzt kommen wir zum generalen Haushalt, allgemeinen Haushalt. Wir haben den Abänderungsantrag 1. Ich λοιπόν, γενικός προπολογισμός και έχουμε την ε, τροπολογία υπαριθμών 1 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. 55 υπέρ. Μία ψήφο κατά και συγχαρητήρια Γιούτα Χάουκ. Τώρα πάμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος με μία τροπολογία υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται και πάμε στην τελική ψηφοφορία αμέσως. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 57 υπέρ, μία αποχή και συγχαρητήρια Γιούτα Και τώρα. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία για τον οργανισμό φαρμάκων με την τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται υπαριθμών 2 τροπολογία σε τμήματα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα και τώρα πάμε στο δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 3, με προφορική τροπολογία, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στην 3, τελευταία φράση, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτωτο. Και τώρα το σημείο 4 παρακαλώ, η τροπολογία 4 υπέρ, κατά. Αποχές. Ε, είμαστε ακόμα σε ψηφοφορίες κύριε μου, δεν έχουμε το δεν να σταματήσω. Απορρίπτεται λοιπόν πιο πολλές οι ψήφοι κατά. Παρακαλώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια νέα πρόταση παρακαλώ σχετικά με την προφορική μου τροπολογία. Μπορώ να σας διαβάσω το κείμενο. Η πρόταση λοιπόν έχει ως εξής. Εάν η εσωτερική υπηρεσία ελέγχου στην ε, έκθεσή της του Σεπτεμβρίου 2010 εξακολουθεί να κάνει την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων, ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΜΑ θα πρέπει να δημοσιεύει ένα κατάλογο όλων των ε, προϊόντων που επιτρέπονται και να αναθεωρήσει την θέση. Αυτή είναι η πρότασή μου. Καλώς, λοιπόν. Η συγγήτρια πρώτα να μιλήσει και η ο υπεύθυνο ε, επικοινωνία. Εγώ μπορώ να το δεχθώ, λέει η κυρία Χάουκ. Μπορούμε να το ψηφίσουμε με την τροπολογία αυτή. Καλώ. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα η τροπολογία υπαριθμών 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη, ο πρόεδρος απερίφθη η 6. Απερίφθη. 7 με προφορική τροπολογία. Και δύο τμήματα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. «59 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στη Ιούτα Χάουκ. So, jetzt kommen wir zur EFSA. Ich habe Και τώρα περνάμε στην ΕΦΣΑ. Ασφάλεια τροφίμων. Δύο τμήματα στην πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το αρχικό κομμάτι τώρα, στο δεύτερο, η αρχή διατύπωση στο δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να το υπερηθεύσουμε, μάλιστα. Καλώς. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα χωρίς προφορική τροπολογία. Το αρχικό κείμενο δηλαδή. Το αρχικό κείμενο της τροπολογίας, όχι του αρχικού κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 13 υπέρ. 47 κατά. Καμία εποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Kommen wir zum Abänderungsantrag 3 mit einem mündlichen. Τροπολογία 3 με προφορική τροπολογία. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 6 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 με προφορική τροπολογία της εισηγητρίας υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά σε παληθεύσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. πέρα. 47 υπέρ. 13 κατά. Εγκρίθηκε βέβαια. Τελική ψηφοφορία τώρα. Άρχεται. Πέρας. 51 ψήφι υπέρ, 10 ψήφι κατά. Και συγχαρητήρια και πάλι στην κυρία Χάουκ. Και τώρα για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ECDC, χωρίς τροπολογίες και ως εκ τούτου μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικά την τελική ψηφοφορία ευθύς αμέσως, άρχεται η ψηφοφορία. σοσιαλδημοκράτες έχουν μία περισεβούμενη ψήφο. Κάποιος πρέπει να βγάλει την κάρτα του. Εντάξει, καλά είμαστε τώρα. Πέρας προφορίας, 58 υπέρ, μία ψήφος κατά. Τώρα έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων με δύο τροπολογίες. Την υπαριθμόν ένα πρώτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. δύο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 59. Ναι. Αποχή μία ψήφι κατά μηδέν. Συγχαρητήρια και πάλι. Dann steigen wir gleich ein mit Abänderungsantrag 1. Wer ist dafür? Προφανώ ο πρόεδρο έχει πέρασει το επόμενο κείμενο. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 2 υπέρ. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την δεύτερη τροπολογία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα περιέχει τώρα περισσότερο ψήφο ψηφομένο μέλος. Παρακαλούμε να βγάλει κάποιος την κάρτα του. Πέρασε πληροφορία τώρα. 24 τα ε, υπέρ, 33 τα κατά. Και άρα η δεύτερη τροπολογία απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα τη δεύτερη τροπολογία. Τώρα πάμε στο τρίτο τμήμα τη δεύτερη τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εγκρίνεται. Παράγραφος υπαριθμών 3, τροπολογία υπαριθμών 3, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 36 υπέρ 24 κατά. Τροπολογία 4 τώρα πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 5. Δεύτερο τμήμα. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, τροπολογία 5, τμήμα δεύτερο. Der Wahlgang ist geschlossen. Ist klar ότι απερίφθη. Ε, Απογοήτευση. 52 ε, κατά. Με 7 ψήφους υπέρ, απερίφθη λοιπόν. Και πάμε στην τροπολογία τρία και την τέσσερα μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχή εγκρίνονται έξι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επτά υπέρ κατά αποχές, αλλά ας επαληθεύσουμε την 7. Πέρας. 23 υπέρ, 36 κατά και απορρίπτεται. Η υπαριθμόν 7. Η υπαριθμόν 8 τώρα. Με προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται υπαριθμόν 9 τώρα προφορική τροπολογία υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται στη 10 υπέρ κατά. Ας επαληθεύσουμε, δεν ήταν σαφές. Επαληθεύουμε λοιπόν τη 10 ηλεκτρονικά. Πέρας. 23 υπέρ, 37 κατά, απορρίπτεται. Και περνούμε στην τροπολογία υπερθυμών 11 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στη 12 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται. Πάμε στα 13 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται προφανώς. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πάμε στο 16 με προφορική τροπολογία. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές και εγκρίνεται. Περνάμε στη τελική ψηφοφορία παρακαλώ. Ηλεκτρονικά και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 57 υπέρ 3 κατά και συγχαρητήρια στον κύριο εισηγητή. Έτσι ολοκληρώνουμε, λέει ο Πρόεδρος. Σχεδόν, σχεδόν. Σχεδόν, γιατί θα ξέχναγα την τελευταία μας γνωμοδότηση, την υπαριθμόν 14, τελευταία ψηφοφορία. Δεν λησμόνισα τη θηλυκή μου πλευρά, αγαπητοί μου φίλοι. Η συγγήτρια δεν είναι παρούσα σήμερα. Μπορούμε όμως να ψηφίσουμε. Προφορική τροπολογία, συγγνώμη, τροπολογία υπαριθμών 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπαριθμών 2, κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμόν 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μάλλον αλλά ας επαληθεύσουμε την υπαριθμόν 5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 αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 15 τώρα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. μόνο 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 του Μάρτιν Κάλαναν υπέρ. Κατά Αποχές. Mm-hmm. Απορρίπτεται. 19α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19b. Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε, πάμε στην 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ. Να επαληθεύσουμε την 22 ηλεκτρονικά. Πολύ ευχαριστώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Ναι. 29 υπέρ, 30 κατά, αποχές 1 απορρίπτεται και καλό ήταν που το επαληθεύσαμε και προχωρούμε στην 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε για άλλη μια φορά, δεν είναι πολύ προφανές, γιατί κάποιοι συνάδελφοι δεν το χέρι. Η 23 παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Πέρας στις ψηφοφορίες. 44 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εγκρίνεται. Και τώρα ηλεκτρονικά η τελική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρασε τη ψηφοφορία. 47 υπέρ. 7 ψήφοι κατά, 4 εποχέ. Και συγχαρητήρια στην συγκέντρια, στη συντάκτρια. Τι απουσία της. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. Παρακαλώ οι συνάδελφοι που σκοπεύουν να παραμένουν στην αίθουσα, να παραμένουν στην αίθουσα και όποιος θέλει να αποχωρήσει παρακαλώ ησύχως. Τώρα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στη συζήτηση της προφορικής ερώτησης της κυρίας Λίντα Μακέιβαν. Ακόμη δεν έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να μην χάνουμε χρόνο λοιπόν, θα έλεγα ας δώσουμε το λόγο πρώτα στη Λίντα να κάνει την εισαγωγή της, την παρουσίαση του θέματος. Το πρόβλημά μου, πρόεδρο είναι πως η ερώτησή μου είναι προς την Κομισιόν και χρειάζεται να είναι παρούσα η Κομισιόν. Αν δεν είναι παρούσα, θα πρέπει να περιμένουμε. Α, είναι παρούσα. Α, γιατί είπατε ότι λείπει. Ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε, όπως είχαμε προβλέψει το πρόγραμμά μας. Και έχουμε εκπρόσωπο τη Επιτροπή για να απαντήσει την προφορική ερώτηση εκ μέρου τη Επιτροπή. Thank Σας ευχαριστώ. Ονομίζομαι Σαμπίν Μπερινιέ και εργάζομαι στη μονάδα που είναι υπεύθυνη για τη καλλιτικά και ε, Η κυρία Ντεστόρη, την οποία αντικαθιστώ, είναι απούσα λόγω ασθένεια. Ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Μακάβανα για την ερώτησή της. Όπως γνωρίζετε, ο κατασκευαστής των ε, εμφυτευμάτων στήθους ε, χρησιμοποίησε ε, βιομηχανική σιλικόνη διαφορετική από αυτή που είχε δηλώσει στα έγγραφα που απευθύνονταν στην αξιολόγηση συμβατότητας για τα εμφυτεύματα στήθους. Είχε, αντί να χρησιμοποιήσει λοιπόν ιατρικού τύπου σιλικόνη, χρησιμοποίησε βιομηχανικού τύπου. Η Κομισιόν παρακολουθεί την υπόθεση αυτή με μεγάλη προσοχή και βρίσκεται σε στενή επαφή με τα κρατημέλη και πιο συγκεκριμένα με τις γαλλικές και τις γερμανικές αρχές ώστε να πάρει μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς έχει συμβεί. Απαντώντα στην ερώτηση της κυρία Μακάβανα, η κυρία Ντεστόρη ανέφερε ότι οι γαλλικέ αρχές απάντησαν στι αρχές του Ιανουαρίου, ενώ οι γερμανικέ αρχές μας έστειλαν πληροφορίες σε σχέση με την ψευδή αξιολόγηση ε, συμμόρφωσης. Λόγω όμως εκκρεμίους διαδικασίες δεν έχουν δοθεί όλες οι πληροφορίες. Ε, δύο σημαντικά θέματα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση τη απάτη τέτοιου τύπου στα κρατημέλη. Κάποια κράτη-μέλη ε, ε, ε, πρότειναν την αφαίρεση των εμφυτευμάτων μάρκας πιπ όπως η Γαλλία και η Γερμανία, ενώ άλλα κράτη-μέλη σύστησαν να παρακολουθούνται στενά οι γυναίκες που έχουν κάνει τέτοιου είδους εμφυτεύματα και να αποφασίζεται κατά περίπτωση το τι θα γίνει, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα. Τα κράτη-μέλη λοιπόν παρακολουθούν στενά την κατάσταση και λαμβάνουν τα μέτρα που θεωρούν ότι είναι σκόπιμο να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο. Ε, ε, ε, έχουμε ζητήσει γνωμοδότηση από Επιστημονική Επιτροπή για την ασφάλεια αυτών των εφηβητευμάτων στήθους και θα έχουμε το πόρισμα μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου 2012. Το επόμενο θέμα είναι το πώς θα προλάβουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Αυτή η περίπτωση συνέβη ενώ η Κομισιόν προετοιμάζει την αναθεώρηση της νομοθεσίας περί ιατρικών εξαρτημάτων ή εμφυτευμάτων ε, θέλουμε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιες περιπτώσεις όπως τα εμφυτεύματα πίπε στο μέλλον. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον καθορισμό και το, παρακολούθηση των κοινοποιημένων ε, οργανισμών από τις εθνικές αρχές. Θέλουμε να βελτιώσουμε την εποπτεία και την ε, επαγρύπνηση. Αυτό θα γίνει μέσω της αυξημένης συνεργασίας ανάμεσα στις αρμόδιες εθνικές αρχές, ώστε να και, υπάρξει κεντρική αναφορά για τις παρόμοιες περιπτώσεις περιστατικά και να βελτιώσουμε και τα κοινοτικά μέτρα. Τέλο, θέλουμε να βελτιώσουμε την ανιχνευσιμότητα και τι σχετικέ απαιτήσει για τα ιατρικά εξαρτήματα ή παρασκευάσματα μέσω, για παράδειγμα, ενό ε, ενός ενιαίου αριθμού εντοπισμού για συγκεκριμένα τέτοια ε, ε, εξαρτήματα. Βεβαίως ε, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και την ασφάλεια των ιατρικών εμφυτευμάτων μαθαίνοντας από την ε, περίπτωση του εμφυτευμάτων που όπως κάναμε ας πούμε για τα ιατρικά παρασκευάσματα μετά από την υπόθεση με αποφασίσαμε να βελτιώσουμε το, τις δοκιμές που γίνονται για τέτοια εμφυτεύματα έτσι ώστε να αποφευχθούν οι πιθανότητες απάτης ή παράκαμψη του νομοθετικού πλαισίου. Σε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να, να συγκεντρωθούν τα προβλήματα, να εξετάσουμε το τι συνέβη και γιατί. Δεύτερον, να αναλύσουμε την ε, ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα με την περίπτωση του περιστατικού και έπειτα να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό η πρότασή μας, όπως αυτή τη στιγμή ισχύει, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα καθώς και να ε, αποφασίσουμε αν χρειάζονται επιπλέον διατάξεις στην πρότασή μας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι προβλήματα όπως η ε, υπόθεση των εκπαιδευμάτων ΠΥΠΕ θα αποφευθούν στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια των ε, δοκιμών ε, αντοχής θα εξετάσουμε κυρίως τις ελεγκτικές δραστηριότητες των κοινοποιημένων οργανισμών, για παράδειγμα την υποχρέωση προαναγγελθήσας επίσκεψη στον κατασκευαστή ή στην δειγματοληψία. Ε, θα εξετάσουμε λοιπόν τους μηχανισμούς ε, επαγρύπνησης. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μόνο ο κατασκευαστής οφείλει να αναφέρει τα περιστατικά και βεβαίως αυξημένη διεθνή συνεργασία θα υπάρξει, για παράδειγμα στον τομέα των ελέγχων. Πιστεύω πως το σύνολο μέτρων που ήδη προβλέπονται, συνδυασμένα με επιπλέον μέτρα που θεωρούνται ε, απαραίτητα μετά από τις δοκιμές θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του συστήματος και θα εξασφαλίσουν που όμως μόνο ασφαλείς ε, ε, ασφαλή εξαρτήματα θα τοποθετούνται στην ευρωπαϊκή αγορά προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Και τώρα λαμβάνει το λόγο πρώτη η Λίντα Μακάβαν Πολλοί συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Θα πρέπει να περιορίσω λοιπόν το χρόνο ομιλία στα δύο λεπτά. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι μεταδίδεται και η συνεδρίαση από τον κύριο By Satellite. Να γνωρίζετε δηλαδή ότι μαγνητοσκοπείται η συνεδρίαση. Κυρία Λίντα Μακέιβαν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που εξετάζει την υπόθεση αυτή πολύ σοβαρά και πολύ σύντομα η Επιτροπή, γιατί όπως και πολλοί κόσμος σοκαρίστηκα με τα όσα αποκαλύφθηκαν για όλη την υπόθεση αυτή των ιατρικών ε, εξετημάτων. Φυσικά ξεκινήσαμε μια απάτη, μια απάτη θελημένη από πλευρά μια εταιρεία και είναι πολύ δύσκολο κανείς να νομοθετήσει κατά ενός ε, ε, δικήματος και θα πρέπει να επικρατήσει η δικαιοσύνη φυσικά. Ε, έχω όμως να κάνω κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Το πρώτο αφορά την υπόθεση των επιθεωρήσεων. Ένα από τα προβλήματα ήταν ότι αυτή η εταιρεία στη Γαλλία κρυβόταν, έκρυβε μάλλον από τους ελεγκτές το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε βιομηχανική σιλικόνη. Σε αυτή τη νέα σας πρόταση προβλέπονται μη προαναγγελθήσεις επιθεωρήσεις γιατί δεν έχει νόημα νόημα να ειδοποιεί τρει εβδομάδε πριν ότι θα πα να ελέγξει, ώστε να έχει ο άλλο το χρόνο να κρύψει ό,τι απάτε κάνει για τι κουκουλώσει. Το δεύτερο είναι ο συντονισμός με το Υπουργείο Υγείας και Τροφίμων της ΣΥΠΑ. Και είναι αλήθεια, το Food and Drugs Administration, είναι αλήθεια ότι η FDA πριν από κάποια χρόνια έγραψε στον αρμόδιο γαλλικό οργανισμό ενημερώνοντας για τις ανησυχίες του και γιατί οι υπόλοιπες αρχές στην Ευρώπη δεν γνώριζαν τίποτα. Μήπως ε, θα μπορούσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να ε, εποπτεύει καλύτερα και να έχει καλύτερο συντονισμό και για τα ιατρικά εξαρτήματα και έπειτα τα στοιχεία που όσοι λέγονται από τα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η βάση δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να καταγράφει τα προβλήματα ε, και τα ιατρικούς μηχανισμούς, οι εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται. Ε, πώς καταγράφονται όλα αυτά. Και Πώς μπορούμε να δούμε, ας πούμε, για τα εμφυτεύματα σιλικόνης. Και έπειτα για την ανείχνευση μιλήσατε για barcode, για σύστημα ανείχνευσης, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό, αυτοί οι οποίοι τοποθετούν τα εμφυτεύματα να καταγράφουν και να κρατούν αρχαία για οποιοδήποτε εμφύτευμα, ώστε όταν υπάρχει πρόβλημα να μπορούμε να τον ειχνεύσουμε αμέσω, να είναι καταγεγραμμένα στη βάση δεδομένα και αμέσω να εντοπίζονται οι άνθρωποι που έχουν βάλει τέτοιου είδου εμφυτεύματα. Για, στη χώρα μου είναι αδύνατο να ξέρει ποιο έχει βάλει τι εμφύτευμα. Ε, ε, στην, στην, τελευταία αναθεώρηση το ζητήσαμε. Ε, θα, θα περιλάβει κάτι στη νέα οδηγία η Κομισιόν για ένα αρχείο. Ευχαριστούμε Λίντα Μακέβανο. Η Φρανσόα Γκρουστέτ τώρα. Όχι, ο κύριο πρώτα. Αναλαμβάνετε εσεί. Ναι, ζητώ συγγνώμη γιατί την κυρία Γκροστέτα έπρεπε να πάει σε κάποια άλλη συνάντηση, με παρακάλεσε να λάβω εγώ. Είναι λοιπόν γαλλική η εταιρεία που ε, κατασκεύασε αυτά τα εμφυτεύματα, αλλά έχουν διατηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και έτσι είναι πολλές χιλιάδες οι γυναίκες οι οποίες, ε, τις οποίες αφορά αυτό το σκάνδαλο και θα πρέπει να διαρωτηθούμε πώς ε, διατυπώνεται η νομοθεσία για τα ιατρικά παρασκευάσματα και πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο ασφαλή για τις γυναίκες. Ενισχύεται πιστεύω η πρόταση κυρία Μακαΐβαν από τα όσα είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κεντρική σημασία είναι τα προϊόντα, τα ιατρικά παρασκευάσματα ε, που παράγονται στην Ευρώπη να ακολουθούν τους ίδιους αυστηρούς κανόνες με αυτούς που ισχύουν για τα φαρμακευτικά παρασκευάσματα. ειδικά για προϊόντα τα οποία βρίσκονται στο όριο του χαρακτηρισμού μεταξύ φαρμάκου και ιατρικού παρασκευάσματος, θα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε προϊόντα που θα αποκρίνονται στις υψηλότερες προδιαγραφές και με 500, με εκατομμύρια πολίτες που εκπροσωπεί η ευρωπαϊκή αγορά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ασφάλεια του καταναλωτή. Πρέπει λοιπόν σε όλη την Ευρώπη να έχουμε στο δυνατόν πιο υψηλές συνθήκες ασφαλείας και τη σχετική παρακολούθηση, το monitoring δηλαδή, το οποίο θα πρέπει να ισχύει τόσο προκαταβολικά πριν από τη χορήγηση της άδειας αλλά και μετά η εποπτεία της αγοράς, το market surveillance δηλαδή, θα πρέπει επίσης ε, να ε, λειτουργεί διαρκώς σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος για να αποφεύγονται τα προβλήματα. Και βέβαια η ενημέρωση. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πότε σκοπεύει να καταθέσει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ζίμπερ και τώρα ο κύριος Λίσε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Λίντα για την πρωτοβουλία. Είναι πράγματι τραγικό αυτό το περιστατικό ή αυτά τα περιστατικά. Το γεγονό ότι ήδη έχει κάνει την σχετική προπαρασκευαστική δουλειά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση τη νομοθεσία για τα ιατρικά παρασκευάσματα και που θα επιτρέπει και καλύτερο, καλύτερο εξοπλισμό του, καλύτερη δηλαδή ε, θωράκιση των εθνικών υπηρεσιών αλλά και ιδιαίτερα της ε, ε, διαδικασίας εποπτείας και παρακολούθησης αγοράς ήδη είναι ε, θετικά μηνύματα. Υπάρχουν από ό,τι έχουμε μάθει μέχρι στιγμής 60 ε, τουλάχιστον επικίνδυνα εμφυτεύματα της εταιρείας PIP στην κλινική αυτή. Αυτό ε, που έχουν εντοπιστεί, αλλά εντωμεταξύ στην ίδια κλινική έχουν εγχειριστεί περισσότερε από χίλιε γυναίκε, οι οποίε τώρα δεν γνωρίζουν καθώ κλείνει η εταιρεία, ε, εάν βρίσκονται σε κίνδυνο ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και να παρακολουθούμε τι συμβαίνει εκ των υστέρων και να εντοπίζουμε τι φέρνει αποτελέσματα και τι όχι. Μια ιδέα από τη Γερμανία, από γερμανούς εμπειρογνώμενους, θα ήταν να γίνεται όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγού, προμηθευτή δηλαδή ο αναπάντεχος απροειδοποιητός έλεγχος, αλλά και στο επίπεδο της ε, λυπής αλυσίδας προμήθειας του προϊόντος, φερειπίν ε, προκειμένου στην κλινική. Και εκεί θα πρέπει να γίνεται απροειδοποιητό έλεγχο και παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει του σχετικού ε, τι σχετικέ επαληθεύσει για να μας πει εάν μπορεί να περιλάβει την πρόταση αυτή στην οδηγία. Στη νέα οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ροτ Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λυπούμε πάρα πολύ που χρειάστηκε να συζητήσουμε το θέμα των ιατρικών παρασκευασμάτων και λοιπόν μηχανημάτων. Είναι για συζήτηση μόνο λόγω ενός σκανδάλου, γιατί αυτό έπρεπε να το έχουμε από πριν ε, συζητήσει και αντιμετωπίσει, πριν εμφανιστούν τα προβλήματα. Ό,τι ακούστηκε λοιπόν πολύ σωστό είναι, αλλά δεν αλλάζει τίποτε ως προς το γεγονός ότι μπορεί και πάλι να εμφανιστεί αντίστοιχο σκάνδαλο. Είναι δυνατό με την υφιστάμενη νομοθεσία το κράτος μέλος να ορίσει συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένους φορείς οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν τεχνικά δεδομένα. Φερρυπίν στη Γερμανία έχουμε 16 τους φορείς. Ε, ο κάθε ένας από αυτούς τους φορείς θα αποφασίσει σε ποιο παραγωγό θα πάει σε πιο προμηθευτή. Ο Γάλλος μπορεί να πάει φερειπίν στον Πολωνό να κάνει έλεγχο, ο Γερμανός στον Ιταλό και το καθεξής. Και όπως είπε η κυρία Λεκρενιέ, ο παραγωγός αυτών των εμφυτευμάτων σιλικόνης έδωσε ψευδή στοιχεία, δηλαδή ε, δήλωσε ψευδός ότι χρησιμοποιεί ιατρικής ποιότητας σιλικόνη αλλά και, το, και να μην ήταν ψευδή τα στοιχεία, δεν θα μπορούσε η εταιρεία πιστοποίηση, η TÜV της, ε, Ρινανίας να επαληθεύσει το όντι αν είναι σωστή ποιότητα τα εμφυτεύματα. Αυτό ισχύει γενικότερα. Και έτσι έρχονται εμφυτεύματα και άλλα παρασκευάσματα στο σώμα το ανθρώπινο χωρί κάποια επαλήθευση. Ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανεξαρτήτω του συγκεκριμένου σκανδάλου ε, δεδομένου ότι το κύριο πρόβλημά μας είναι οι αρχές επιτήρησης επαλήθευσης. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Μία έστω, ένας φορέας, ε, ε, είτε πρόκειται για, τον, για την Εθνική Αρχή Φαρμάκων, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Αρχή Φαρμάκων του Λονδίνου, πρέπει ένας φορέας να φέρει την ευθύνη για τους ελέγχους. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης, εάν συμφωνεί όπως ε, πιστεύω εγώ ότι χρειάζονται άλλες διαδικασίες αδειοδότησης. Οι κατηγορίες ιατρικών παρασκευασμάτων και μηχανημάτων ε, από την πρώτη έως και την τρίτη ε, χρειάζονται πολύ πιο αυστηρούς ελέγχους. Γιατί αν πάρουμε συνδυασμένα προϊόντα αυτών των τριών κατηγοριών, τότε είναι πολύ πιο ισχυρή η, η, η ουσία Μπορεί να υπάρξουν πολύ πιο επικίνδυνε ουσίε σε συνδυασμό και γι' αυτό χρειάζονται πολύ πιο αυστηρή έλεγχη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Θα πρέπει να κλείσουμε τον κατάλογο των ερωτήσεων. Έχω τον κύριο Chris Davis στον κατάλογο μου, την κυρία Ραβεζή, Πανιό, Αντωνέσκου, Σίλτερ, Σάιντεμο. και πολλούς πολλούς άλλους. Ja, ist mit Όχι, έχω σημειώσει και εσάς. So, dann ist die κλείνει ο κατάλογος των αγορητών. 1,5 λεπτό θα έχετε όμως ο καθένας από εδώ και μπρος. Chris Davis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα για την Κομισιόν τα εφητεύματα στήθους από τη Γαλλία ήταν εγκεκριμένα από το ρυθμιστικό οργανισμό της Γαλλίας και τους είχε δοθεί ε, το σήμα ε, συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε «Ε» και αν ναι, τα εθνικά ρυθμιστικά σώματα, οι οργανισμοί έχουν οποιαδήποτε δυνατότητα να προλάβουν το, διαφήμιση, την εμπορία τέτοιων προϊόντων στις υπόλοιπες χώρες. Als ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να θυμίσω στους συναδέλφους ότι ωστόσο υπήρξαν πάνω από 500.000 ε, γυναίκες που ε, έλαβαν αυτά τα εμφυτεύματα σε ολόκληρο τον κόσμο. 30.000 στη Γαλλία, 30.000 στην Αγγλία, αλλά οι περισσότερες στη Λατινική Αμερική. Όταν μιλάτε ότι υπήρχε πρόβλημα πιστοποίησης και η πιστοποίηση δεν έγινε, όπως είπε ο συνάδελφος, από οργανισμό γαλλικό, αλλά από οργανισμό ε, γερμανικό. Μόνο που αν ο οργανισμός πιστοποιεί, θα πρέπει τη στιγμή που κάνει ελέγχους ε, στο εν λόγω εργαστήριο, δεν θα πρέπει να τους προειδοποιεί, γιατί ο κύριος Μάος που ήταν ο διευθυντής εξαφάνισε όλα τα προϊόντα που έδειχναν ότι αυτό το ζέλ ήταν ε, ε, βιομηχανικό και όχι ιατρικό. Εφόσον είχε υπάρξει πιστοποίηση λοιπόν και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να έχει κανείς το σήμα CE αυτό πρέπει να είναι απροειδοποίητο, ε, πρόσμενο έλεγχο, γιατί διαφορετικά είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου μόλι έχετε κάποιον απαταιώνα, εξαφανίζει όλα τα προβληματικά προϊόντα. Έπειτα, οι εθνικοί οργανισμοί, και αυτό με έχει προβληματίσει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι χειρούργοι τη Μασαλία, μάλιστα, είχαν διαπιστώσει το 2008 ότι υπήρχαν δυσλειτουργίε και είχαν ε, έρθει σε επαφή με τις εθνικές αρχές. Εδώ λοιπόν θα πρέπει οι εθνικές αρχές πιο γρήγορα να ανταποκρίνονται στις παρενέργειες αυτών των εμφυτευμάτων και τρίτο ακόμα που, σημείο που ήθελα να το πω και κανένας δεν το συζητά είναι και η ευθύνη των χειρουργών. Μα πώς γίνεται χειρούργοι εδώ και χρόνια να χρησιμοποιούν αυτά τα εμφυτεύματα, να έχουν την επαφή με τις ε, γυναίκες γιατί ε, έσπαγαν τα εμφυτεύματα και να μην λένε τίποτα. Πώς είναι δυνατόν. Από νομικής άποψης λοιπόν υπάρχει και η ευθύνη των χειρούργων. Μα βγάζουν τρελά λεφτά με τα εμφυτεύματα στήθος οι χειρούργοι. Κυρία συνάδελφε, πρέπει λοιπόν να υπάρχει τέτοια νομοθεσία και πρέπει και αυτοί να φέρουν την ευθύνη τους. Και έπειτα έχουμε ένα πρόβλημα με το vaginal mesh. Και θα ήθελα στο... στο θέμα των δοκιμών αντοχής να μας πείτε τι συμβαίνει με αυτά τα vaginal mesh. Ναι, ευχαριστώ παρακαλώ. Να είσαι ώστε να τον πιο σύντομη για να είμαστε δικοί προς όλους τους συναδέλφους. Για να προλάβουν όλα, να μιλήσουμε κύριο Σπανιό. Αλλά πώς το λέω. Ευχαριστώ. Διαπιστώνουμε συλλογικά ότι εκ νέου βρισκόμαστε σε ένα σκάνδαλο υγειονομικής ασφάλειας στην Ευρώπη, όπως έγινε επίσης με το Mediator. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια απάντηση. Μετά από επιθεώρηση, από έλεγχο, είδαμε ε, ε έλεγχο στο εργοστάσιο, έγινε ο εντοπισμός ε, ελαττωματικών εμφυτευμάτων εκεί. Έπειτα υπάρχει επιβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνώριζε το 2005 και το 2006 κατατέθηκαν πολλές καταγγελίες στη Μεγάλη Βρετανία, στη Μεγάλη Βρετανία ε, κατά της ΠΕΙΠ και στην Γαλλία το ίδιο και ότι οι Γάλλοι ε, πλαστικοί χειρούργοι ματέως προσπάθησαν να προσελκύσουν την προσοχή των αρμόδιων γαλλικών οργανισμών το 2008-2009 ναι, ξέρουμε τώρα πως αυτή η εταιρεία έχει τεθεί υπό ε, νομικό έλεγχο και έχει κηρύξει πτώχευση και ότι ήταν πολύ φθηνότερα όλα αυτά τα επιτεύγματα από ότι τα άλλα. Και εδώ δεν έχουμε απαντήσεις. Ε, εδώ υπάρχουν, όπως το θύμισε και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει μια οδηγία που υπήρχε. Υπήρξε λοιπόν παράβαση που διαπιστώθηκε σε σχέση με αυτήν την οδηγία. Αν και, και εδώ σας δικαιολογώ ότι θα πρέπει πρέπει τώρα να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρξει βελτίωση της εν λόγω οδηγίας μέσα στο πλαίσιο των όσων προετοιμάζονται για τα ιατρικά σκευάσματα. Κυρία Αντωνέσκου και παρακαλώ 1,5 λεπτό αυστηρά. Ε, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι η υπόθεση για την οποία μιλάμε σήμερα έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα σε σχέση με την ασφάλεια και την ανάγκη ρύθμισης. Ωστόσο, εδώ και καιρό γίνεται λόγος για αυτό το είδους την ανάγκη βελτίωσης ε, της ε, σχετικής νομοθεσίας και γι' αυτό θέλω να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη νέες τεχνολογίες και η πρόοδος της τεχνολογίας, όπως η νανοτεχνολογία για παράδειγμα. Χρειάζεται νομοθεσία πολύ πιο αυστηρή κατά τη γνώμη μου όσον αφορά αυτή την τρίτη κατηγορία διατάξεων συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εποπτεία και καλύτερη ανεχνευσιμότητα για τα εμφυτεύματα, αλλά χρειαζόμαστε και μια ενημέρωση από πλευράς των καταναλωτών και καλύτερη ενημέρωση των συνδέσμων καταναλωτών. Έχουμε τώρα 80 οργανισ... κοινοποιημένους οργανισμούς. Χρειάζεται διαρκώς να χρησι... μάλλον χρειάζεται να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Περιμένουμε από πλευρά της Κομισιόν καλύτερη νομοθεσία, πιο διαφανή. Ε, όμως σεβόμενοι τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ, Σάρλες. Uh, um, Ευχαριστώ. κυρία Childers. Συμφωνώ και εγώ με τις άλλες ερωτήσεις, αλλά έχω και μία ακόμα, περισσότερο μία προειδοποίηση, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν λαμβάνει η χώρα ένα τέτοιο γεγονός, καλό είναι να έχουμε μία ιατρική ανάλυση για το πώς ε, συνέβη αυτό που συνέβη κατά πρώτο λόγο. Πρώτα δηλαδή να το αναλύσουμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το συμβάν αυτό και να αποφύγουμε νέους κινδύνους. Όσον αφορά τώρα τον έλεγχο των ε, οργάνων που κοινοποιούν και εγκρίνουν και όσον αφορά τον έλεγχο, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ή μεταχείριση σε όλες τις χώρες. Στη δικιά μου, για παράδειγμα, τα όργανα αυτά, τα σώματα αυτά, ε, την κάνουν ε, τη δουλειά αυτή και μερικές φορές ε, την κάνουν, αλλά υπάρχει και επικάλυψη με άλλα όργανα. Μήπως λοιπόν πρέπει να δούμε ποιος κάνει αυτή τη δουλειά στην κάθε χώρα και να φροντίσουμε να μην υπάρχει υπερβολική, υπερβολικός ζήλος από ένα σώμα όταν υπάρχει και κάποιο άλλο σώμα στην ίδια χώρα ή σε κάποια άλλη χώρα που κάνει την ίδια δουλειά. Να μην υπάρχει επικάλυψη λοιπόν στους ελέγχους και στα σώματα τα οποία κοινοποιούν τις άδειε. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Σαλτεμός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Υπάρχει πρόβλημα εδώ, οπότε ρωτάω την Επιτροπή. Ευρωπαίοι ασθενεί πότε θα μπορέσουν να έχουν εμπιστοσύνη στα φυτέυματα που δέχονται. Ακούσαμε ότι 500 περίπου ε, πήραν ε, τεχνητό μυρό και πέρυσι η εταιρεία απέσυρε το προϊόν αυτό. Άρα, ορισμένοι ασθενείς σήμερα δεν ξέρουν πότε θα αντικατασταθεί ο μυρός αυτός. Συνεπώς, Ούτε η έρευνα στην αγορά είναι αρκετά καλή. Ούτε ασφάλεια των προϊόντων ε, έχουμε με σιγουριά. Καταλαβαίνετε ότι οι Ευρωπαίοι ασθενείς πρέπει να ξέρουν ότι μπορούν να εμπιστεύονται τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Καλό λοιπόν θα είναι να ξέρουν πότε θα γίνει αυτό και πότε θα υπάρχει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για τον έλεγχο και την εποπτεία. Ευχαριστούμε. Τώρα η Σοφία Κόνη έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλά υπόθηκαν ήδη. Τρία σημεία έχω εγώ να θίξω μόνο. Πρώτον, αυτά τα ιατρικά εμφυτεύματα είναι ε, τέτοια που να βοηθούν τους ασθενείς. Είτε πρόκειται για τα εμφυτεύματα, είτε πρόκειται και για άλλα εξαρτήματα που μπορεί να είναι οι βηματοδότε ή άλλα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούν προσωρινά ή σε μόνιμη βάση ασθενεί. Δεν απαιτούν ε, κάποια διαδικασία όπως γίνεται με τα φάρμακα για να μπουν στην αγορά και να διατεθούν στην αγορά. Οπότε ρωτάω και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως θα έπρεπε να προβλέψουμε μια διαδικασία και για τα εξαρτήματα αυτά που να είναι εξίσου λεπτομερεί όπως εκείνη που ακολουθούμε για τη διάθεση στην αγορά των φαρμάκων. Έπειτα η εταιρεία η οποία έκανε την απάτη, λέει ότι πήρε την άδεια από ένα γερμανικό εργαστήριο για τα φυτέυματα αυτά, γιατί το γερμανικό εργαστήριο ήταν πιο ελαστικό από ό,τι άλλα γαλλικά ή βέλγικα αντίστοιχα. Μήπως λοιπόν και εδώ θα έπρεπε να προβλέψουμε, και απευθύνομαι στην Κομισιόν εδώ, Μήπως έπρεπε να προβλέψουμε εναρμόνιση των ελέγχων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε ένας Γάλλος επιχειρηματίας να μην μπορεί να διευκολύνει εντό αγωγικών τις διαδικασίες και να παίρνει πιο εύκολα μια άδεια από ένα γερμανικό εργαστήριο. Και έπειτα για τις άδειες. Όταν πάμε σε ένα εστιατόριο να ελέγξουμε αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, κάνουμε ελέγχους χωρίς να προειδοποιήσουμε. Ευτυχώς, εννοείται. Πώς είναι δυνατόν εδώ τώρα να ειδοποιούμε ότι θα πάμε να ελέγξουμε. Μα δεν είναι τις βιομηχανίες που πρέπει να διευκολύνουμε για να προστατεύσουμε, αλλά τους καταναλωτές, τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Η Γιολάντα Αγίπνερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, τώρα ασχολούμαστε με μια πολύ δύσκολη περίπτωση μία περίπτωση που έχει να κάνει με την ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις γυναίκες αυτή τη φορά, οι γυναίκες οι οποίες αναρώνουν από καρκίνο ή από κάτι άλλο και χρησιμοποιούν τέτοια φυτέυματα σιλικόνης. Ρωτάω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι σκοπεύει να κάνει όσον αφορά τους ελέγχους από πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πληροφορία για την απειλή αυτή στην υγεία των γυναικών που έχουν λάβει τέτοια φυτεύματα και πότε ξεκίνησε τους ελέγχους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπετε, δεν θέλω εδώ να τα βάλω με το ιατρικό προσωπικό που χρησιμοποιεί τέτοια εμφυτεύματα και τα δίνει στις γυναίκες αν είχαν πάρει την άδεια όπως πρέπει, τότε λογικό είναι να τα χρησιμοποιούν. Δεν πρέπει πάντα να σκέφτονται «Α, κάτι δεν πάει καλά, πώς να το σκεφτούν αυτό». Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει ώστε να επιστήσει την προσοχή και άλλων εταιριών για το ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τέτοια κακά υλικά. Ευχαριστώ. Κύριε Βάσκεβα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι βέβαια ιδιαίτερα εγκληματική η ενέργεια που προκάλεσε το σκάνδαλο στη Γαλλία με τα εμφυτεύματα στήθους, αλλά θα πρέπει γενικότερα να μεριμνήσουμε να ενισχυθούν περισσότερο οι έλεγχοι ποιότητας με τη νέα οδηγία. Δεν είναι δυνατόν εμφυτεύματα στήθους τα οποία έχουν, στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί σιλικόνη για στρώματα αντί για ιατρικού τύπου σιλικόνη να φτάνουν μέχρι τις αγορές ε, και τα χειρουργεία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται έγκαιροι και σωστοί έλεγχοι για να αποτρέπονται τέτοιου είδους περιστατικά. Αλλά θα διαφωνήσω με την κυρία Ροτπέρεντ η οποία είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφορετικό σύστημα για την αδειοδότηση και ότι δεν χρειάζονται οι ε, έλεγχοι, οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Δεν συμφωνώ σε αυτό γιατί μπορεί να υπάρξουν ε, παραποιήσεις ή να υπάρξει διάθεση προϊόντων ε, με ανεπαρκή ποιότητα στην αγορά και γι' αυτό πρέπει να είμαστε παρόντες και να ελέγχουμε όχι μόνο στην παραγωγή του προϊόντος αλλά και όπως είπε ο κ. Πέτερλής μέχρι το σημείο όπου γίνεται η εμφύτευση στον ασθενή. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα του ελέγχου και της επαλήθευσης ώστε να αποφεύγουμε και τις ε, παραποιήσεις ή ε, απομιμήσεις προϊόντων σε αυτό είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι χρειάζεται να γίνονται οι έλεγχοι και βέβαια η επαλήθευση του Εθνικού Μητρώου. Ευχαριστώ κυρία Κούκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Τα ιατρικά εξαρτήματα, μεταξύ άλλων και τα εμφυτεύματα, σε ένα μεγάλο βαθμό αποτελούν και πηγή εσόδων και κέρδους. Και πολλές φορές χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν είναι διαφανής ο ιατρικός προϋπολογισμός. Φυσικά και υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τέτοια εμφυτεύματα επειδή έχουν περάσει από καρκίνο του στήθους. Όμως οι γυναίκες πρέπει να σκέφτονται διαφορετικά. Πρέπει οι νομοθεσία να περιλαμβάνει την υποχρέωση για καλύτερη ενημέρωση, για πληροφορίες και να μάθουν οι γυναίκες ότι το μέλλον και η μόδα δεν είναι ε, το στήθος με σιλικόνη, αλλά η υγεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε και οι γυναίκες έτσι να αλλάξουν κάπως νοοτροπία. Πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό στην πρόταση για νομοθεσία. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνος τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο πράγματα έχουμε εδώ. Το ένα είναι τι κάναμε όταν ανακαλύψαμε το πρόβλημα, κάτι το οποίο έκανε πιο μεγάλους ακόμα τους φόβους των γυναικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, οι Βρετανικές αρχές αντέδρασαν εντελώ διαφορετικά από τις Ιρλανδικές αρχές. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Όπως έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και έχουμε καλό συντονισμό όσον αφορά την αντίδρασή μας εφόσον υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα ιατρικά εξαρτήματα. Έτσι ώστε να μπορούμε να καθησυχάσουμε τους ε, ασθενείς. Τώρα σε ορισμένες χώρες ε, μέλη οι πολίτες, οι ασθενείς είναι τρομαγμένοι και σε άλλε όχι, εκεί που τους λένε ότι δεν πρέπει να αφαιρέσουν, δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Είναι τελείως διαφορετική δηλαδή η πληροφορία που παίρνουν και άρα και οι φόβοι των ε, γυναικών. Δεύτερον, υπήρξε απάτη. Αυτό είναι σαφές. Οι έλεγχοι όμω πρέπει να πάνε πίσω. Νομίζω ότι οι προμηθευτέ αυτή τη βιομηχανική σιλικόνη πρέπει να ελεγχθούν για το πού έστειλαν το προϊόν τους αυτό. Και εδώ πρέπει να αναλάβουμε δράση. Διότι θα ζήσουν περισσότερο. Εδώ πέρα μιλάμε για τα εμφυτεύματα στήθους, αλλά υπάρχουν και άλλου είδους εμφυτεύματα. Αναφέρθηκαν σε αυτά οι συνάδελφοι. Όπως είπε και κάποιος συνάδελφος, υπήρξε πρόβλημα και με κάποιους τεχνητούς μυρούς. τεχνητούς γλωτούς. Και νομίζω ότι και εκεί πρέπει να πάμε πίσω και να ψάξουμε πώς ε, έχει προχωρήσει το πράγμα. Ροντρίγιος τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο θέμα εδώ και αυτό είναι ότι στα κράτη-μέλη φτάνουν προϊόντα τα οποία δεν είναι καλά. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το ψάξει σε βάθος και να ε, αποφασίσει ποιο έχει την ευθύνη. Διότι οι άδειε που δίνουμε δεν πρέπει να είναι γραφειοκρατικές καθαρά. Πρέπει να ξέρουμε ότι όντω γίνονται έλεγχοι, χωρίς προειδοποίηση φυσικά, δεν μπορεί να προειδοποιούμε ότι θα πάμε να ελέγξουμε και να παρακολουθούμε και τα προϊόντα αυτά. Επειδή ακριβώ δεν τα είχαμε αυτά, γι' αυτό καταλήξαμε σε αυτό το σκάνδαλο με κεφαλαίο σίγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει συστάσει στι χώρε μέλη. Εγώ συμφωνώ ότι οι χώρε μέλη είναι κυρίαρχε, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση ε, στι γυναίκε ανάλογα με το από ποια χώρα προέρχονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, αν μη τι άλλο, να κάνει συστάσει έτσι ώστε όλε οι γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Δεν χρειαζόμαστε νέους κανόνες, πρέπει να διορθώσουμε όμως ότι δεν πάει καλά μέχρι τώρα. Εδώ δεν υπήρχαν έλεγχοι και άρα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί οι οποίοι έσφαλαν και δεν φρόντισαν να γίνουν οι έλεγχοι αυτοί. Κάποιος ε, μπορεί να χρησιμοποιεί κάποια προϊόντα, το οποίο κατά 25% να είναι καλά, κατά 70% όχι. Ε, πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να κάνουν συστάσεις τα κράτη-μέλη πάνω απ' όλα για να μην υπάρχει ανισότητα μεταξύ των γυναικών. Μάριο Πιρέλη τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Λίντα που μας έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αυτή η γαλλική εταιρεία, η PIP, που κατασκεύασε αυτά τα λατωματικά εμφυτεύματα, φέρει τεράστια ευθύνη απέναντι στην ανθρωπότητα. Στην Ιταλία έχουν γίνει πολλές καταγγελίες ε, στη δικαιοσύνη, γιατί αυτό το εμφύτευμα μπορεί να προκαλέσει όγκο στο μαστό. Στη Γαλλία σκέφτηκαν να αφαιρέσουν ε, γύρω στις 30.000 ελαττωματικά εμφυτεύματα. Αλλά αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι αυτή η γαλλική εταιρεία έχει εξάγει το 80% της παραγωγής της στην Ευρώπη και στην Λατινική Αμερική. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να μας κάνει να τα σκεφτούμε. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη επαφή ανάμεσα στα κράτη-μέλη και καθημερινά να γίνονται έλεγχοι. Νομίζω πως αυτό πρέπει να γίνει και η Κομισιόν θα πρέπει να το προσέξει πολύ αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Και τώρα η Ελιζαμπέτα Γκαρδίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω πως πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσουμε την ανιχνευσιμότητα των εξαρτημάτων, ότι πρέπει να ορίσουμε κριτήρια για τους οργανισμούς κοινοποίησης για να μπορούμε να εγγυηθούμε την αυστηρότητα και την ανεξαρτησία των οργανισμών και να έχουμε και ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης των κινδύνων θα ήθελα να εκμεταλλευτούμε τα όσα αποκαλύφθηκαν με αυτή την υπόθεση για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στις γυναίκες, να τους εγγυηθούμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Εγώ συζητώντας με γιατρούς, ακτινολόγους στην Ιταλία, άκουσα από αυτούς και μου το επιβεβαίωσαν ότι οποιαδήποτε και αν είναι το εμφύτευμα στο στήθος αποτελεί, ακόμα και αν γίνει με βάση όλα τα κριτήρια, αποτελεί ένα εμπόδιο στην πρόληψη του καρκίνου, διότι εμποδίζει την ε, ε, όραση στην περιοχή αυτή. Δηλαδή εμποδίζει τις ε, ακτίνες. Και αυτό πρέπει να το πούμε στις ε, γυναίκες ε, και πρέπει να λάβουμε υπόψη πως νεότατες κοπέλες ε, κάνουν τέτοιου είδους εγχειρήσεις με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγει το σκίνδυνο. Και έπειτα να ρωτήσω τα όσα έμαθα ε, είναι αλήθεια ότι δηλαδή φαίνεται πως ο εφευρέτης των εφητευμάτων Πίπε προσπαθεί να συνεχίσει τη δουλειά του με άλλο όνομα. Έχει ε, φτιάξει μια άλλη εταιρεία με, ε, με, με τους γιους του, στο όνομα των γιών του και ετοιμάζεται να φτιάξει 400 εφητεύματα ημερησίως. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα την Γενική Διευθύντρια της Γενικής ε, η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διευθύνσεως ε, Προστασίας του Καταναλωτή και της Δημόσιας Υγείας είναι εδώ. Παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τη νέα πρόταση. Η κυρία Ροντμπέρεν, η Λίντα Μακέβιν, ο Πίτερ Λίζε μας ρωτάνε τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Ε, λοιπόν, όπως ε, λένε και οι συνάδελφοι, θα κάνουμε αυτό που ονομάζουμε stress test. Δηλαδή, αναλύουμε τη δικιά μας πρόταση, η οποία ήταν ε, ήδη έτοιμη, προκειμένου να δούμε κατά πόσο αυτό που προτείνουμε θα μπορέσει να αποφύγει τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον, σαν και αυτήν που αντιμετωπίσαμε πρόσφατα. Προς το παρόν, πρόθεσή μας είναι να ενισχύσουμε και να κάνουμε πιο αυστηρούς τους ελέγχους στην αγορά και την ανεχνησιμότητα. Όμως δεν σκεφτόμαστε να ακολουθήσουμε και την ε, οδό που μιλάει για άδειε ε, πριν τη διάθεση στην αγορά. Θέλουμε να φροντίσουμε όλες οι εθνικές αρχές να έχουν εξίσου τη δυνατότητα ελέγχων δεν είναι θέμα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να έχει κανείς την επιλογή να πάει στο ένα εργαστήριο, στο ένα σώμα ή στο άλλο σώμα. Όχι. Τα σώματα εκείνα τα οποία έχουν οριστεί και είναι αρμόδια για τους ελέγχους, αυτά τα σώματα θα πρέπει να δρουν όλα στο ίδιο επίπεδο, με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες μέλη. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να φροντίσουμε αυτή η δυνατότητα ελέγχου να υπάρχει με τον ίδιο τρόπο και να υπάρχει διαφάνεια στους ελέγχους αυτούς που φέρουν σε πέρα στα κράτη-μέλη. Να γίνεται ο ίδιος έλεγχος δηλαδή σε όλες τις χώρες. Έπειτα, όπως είπε η κυρία Μακάβεν, οι έλεγχοι δεν πρέπει να γίνονται μετά από προειδοποίηση ενημέρωση της βιομηχανίας. Όχι. Και έτσι κι αλλιώς ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο της παραγωγής μέχρι το επίπεδο των ασθενών. Και τρίτον, χρειαζόμαστε την ανεχνευσιμότητα. Όπως λέει και ο Πίτερ Λίζε, δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι γυναίκες στις οποίες μπήκαν τα εμφυτεύματα αυτά. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος ε, για να εντοπίσουμε τα εμφυτεύματα αυτά και έτσι να ξέρουμε ε, σε ποιους ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και μια βάση δεδομένων πλήρη. Προς το παρόν έχουμε μία αλλά δεν είναι πλήρης. Έτσι ώστε να μπορούμε να ανοιχνεύουμε ε, την ε, κατάσταση σε όλη την αλυσίδα από την παραγωγή μέχρι τον ασθενή. Έπειτα το θέμα δεν είναι το θέμα της ε, άδεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έφταιγε η άδεια. Το πρόβλημα ήταν ο έλεγχος, η εποπτεία της αγοράς και η παρακολούθηση της ανεχνευσιμότητας. Τώρα πολλοί συνάδελφοι ρωτάουν γιατί φτάσαμε εκεί. Η αλήθεια είναι ότι το FDA έκανε ελέγχους κατά το παρελθόν. Δυστυχώς πρέπει να σας πω την αλήθεια ότι το FDA έκανε το 2000 τους ελέγχους αυτούς των εφητευμάτων δηλαδή, όχι για τη σιλικόνη, αλλά για τα άλλα ποσά line. Και η FDA απέσυρε την άδεια, δεν επέτρεψε δηλαδή τα προϊόντα αυτά της συγκεκριμένη εταιρεία που ήλεγξε, τα σταμάτησε, δεν τα άφηνε να εισαχθούν πια. Εμείς δυστυχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε δεν ενημερωθήκαμε. Τώρα ενημερωθήκαμε. Και τώρα, αρχές Ιανουαρίου, 10 Ιανουαρίου, μας δώσανε την ε, απάντηση στην ερώτησή μας με τις πληροφορίες που ζητούσαμε. Αλλά αυτές τις πληροφορίες δεν τις είχαμε πριν. Δυστυχώς, γιατί αν είχαμε αυτή την πληροφορία νωρίτερα, θα μπορούσαμε να είχαμε παρεύει και νωρίτερα. Και γιατί δεν την είχαμε αυτή την πληροφορία πριν. Είναι βέβαια απόρριτες οι πληροφορίες αυτές και εμείς έχουμε συμφωνία με τις νομολιτίες από το 2007 για το απόρριτο. Η συμφωνία αυτή φυσικά ισχύει για ό,τι γίνεται μετά το 2007, όχι για το τι γίνεται πριν. Έπειτα, τι πρέπει να κάνει η αρμόδια αρχή βάσει της σημερινής νομοθεσίας και απαντά στον Chris Davis. Οι αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι μόνο προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τους κανόνες διατίθεται στην αγορά. Δηλαδή υπήρξε υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις και για τις γαλλικές βάσει της εποπτείας της αγοράς να διασφαλίζουν ότι μόνο ε, συμμορφούμενα με τους κανόνες προϊόντα διατίθεται στην αγορά. Και ε, μπορούν οι αρχές των χωρών να απαγορεύσουν τα προϊόντα. Το Μάρτιο του 2010 λοιπόν όταν είχαμε το πρώτο ε, σήμα που έλεγε ότι υπήρξε ενδεχομένω πρόβλημα ε, που συνδέεται με τον καρκίνο από τα φυτεύματα αυτά, τότε σταμάτησε η άδεια. Θέλω να απαντήσω και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις στην κυρία Ριβάζη όσον αφορά αυτά τα κολπικά εμφυτεύματα. Νομίζω ότι ναι, και εδώ πρόκειται να... ότι πρέπει να συνεχίσουμε ε, να ενημερωνόμαστε. Δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει όμως. Είναι αλήθεια ότι 80-90% ε, των ε, ευνετεμάτων αυτών εξάγονται. Ένα μικρό κομμάτι των προϊόντων αυτών είναι στις χώρες μας. Εμείς συνεργαζόμαστε σε διεθνές επίπεδο με τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία και προσπαθούμε τώρα να αναπτύξουμε μια νομική βάση ώστε να μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες μετά από ελέγχου που γίνονται σε διεθνές επίπεδο. Αλλά σας λέω πρόκειται για πληροφορίες που είναι απόρριτες και δεν είναι δυνατόν αυτή η ανταλλαγή ε, πληροφοριών να γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Το προσπαθούμε όμως γιατί για μας είναι αναγκαίο. Πότε θα έχουμε την νέα μας πρόταση. Τον Μάρτιο προβλέπετε. Ίσως καθυστερήσουμε λίγες εβδομάδες γιατί η Επιτροπή μου θέλει να φροντίσει αυτή η πρόταση να είναι τέτοια που να αποφεύγονται αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον. Και να ξέρετε ότι θα είσαστε ενήμεροι. Μόλις έχουμε ολοκληρώσει ε, αυτό το stress test που σας είπα στην αρχή, θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τεστόρη. Η Λίντα Μακέβαν παρακαλώ να λάβει το λόγο. Βλέπω πως η κυρία Ροτ Μπέρεν θέλει να κάνει υπερώτηση. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις διευκρινήσεις. Πολλά από τα όσα ρωτήσαμε τα εξετάζει η Κομισιόν. Αλλά θέλουμε να δούμε τα όσα μας είπε η κυρία Ντιστόρη για τη νέα νομοθεσία. Απλά θέλω να ρωτήσω όμως... Ε, το Ευρωπαϊκό Οργανισμός Φαρμάκων είναι ε, το αντίστοιχο του FDA. Δηλαδή τι το FDA πάει στην Γαλλία ερευνά και κανένας δεν ξέρει ξέρει τίποτα για όλα αυτά. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο επαφής και ε, βάση δεδομένων ε, να έχουμε τη δυνατότητα στην Ευρώπη να το κάνουμε αυτό. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον οργανισμό που ήδη υπάρχει στο Λονδίνο. Α, τώρα, αν οι κυβερνήσεις θέλουν να κρατήσουν το αρμοδιότητές τους, μα η ασφάλεια των ασθενών είναι πρώτη, προηγείται. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω ξαναρχίσει να ξανανοίξουμε το γύρο των ερωτήσεων. Γι' αυτό παρακαλώ να περιοριστούμε μόνο σε συζήτηση μεταξύ των συντονιστών. Να το αφήσουμε δηλαδή για τους συντονιστές. Είναι ένα θέμα που χρειάζεται περαιτέρω. Μελέτη ούτως ή άλλως. Κύριε Μπέρεντ, πρόεδρε, στα αγγλικά. Δεν θέλω να κάνω τη δύσκολη και ξέρω ότι είμαι η κακιά, αλλά νομίζω ότι η κυρία Στόρη θα πρέπει να πάρει και το μήνυμα από εμά όταν φύγει και όχι να το κάνουμε, να συζητήσουμε το θέμα μεταξύ συντονιστών, γιατί η κυρία Στόρη πολύ καλά τα είπε, ο συνήθως ε, κατά 90%, αλλά το 10% που δεν μας απαντά ικανοποιητικά είναι το τι κάνουμε από εδώ και μπρος και τέτοια, τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν τέσσερις τάξεις, τέσσερις κατηγορίες δηλαδή ιατρικών παρασκευασμάτων. 1, 2α, 2β, 2γ. Και μάλλον 2α, 2β και 3. Και πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξει η σχετική νομοθεσία. Λέτε ότι, δε, ότι χρειάζεται νομοθεσία ή μάλλον διαδικασία για την αδειοδότηση. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ε, ίσως όχι για την πρώτη κατηγορία, αλλά για τις άλλες ναι. Αλλά πάντως πρέπει να έχουμε και σαφείς ορισμούς. Ε, ο χρόνος δρά αντίθετα με εμάς. Δηλαδή θα προχωρούν πολύ γρήγορα τα νέα ιατρικά παρασκευάσματα που θα βγαίνουν στην αγορά και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε τι εξελίξει. Και Πρόεδρε, ξέρω ότι η πρώτη μέρα που έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σα δεν πρέπει να κάνω την κακιά, θα προσπαθήσω να το αποφύγω στο μέλλον, αλλά πρέπει να προλάβουμε το τρένο, όπω είπε και η κυρία Μακέιβαν, πρέπει να είμαστε εμεί η μηχανή, ο, ο που θα φέρνει το τρένο αυτό μπροστά, να μην περιμένουμε από τα κράτη-μέλη και πρέπει να οργανωθούμε κάπως καλύτερα. Είναι κακές οι επιδόσεις των οργάνων κοινοποίηση, των φορέων κοινοποίηση στα κράτη-βέλη. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη λοιπόν αυτό και να δράσουμε αναλόγω. Ο κύριο Χρότε. Ναι, τώρα συμβαίνει αυτό το οποίο φοβόμουν. Να δίνω το λόγο σε έναν και τον ζητούν όλοι. 30 δευτερόλεπτα από τον κύριο Σπαγιό, αλλά κλείνει ο κατάλογο γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Να πω μόνο ότι δεν απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις, κυρία εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρίσκω το, να μην απαντάτε στις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στη Γαλλία το 2005-2006 σημαίνει ότι και εκεί υπήρξε μια πλήρης παραπληροφόρηση ή μη πληροφόρηση και τίποτα μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπόρεσε να γίνει. Άρα λοιπόν φέτο, ε, τώρα πρέπει να εξετάσουμε εμείς οι ευρωβουλευτές αν δεν υπήρξε παράβαση της οδηγίας όπως ισχύει σήμερα ή μήπως ε, δεν ε, ε, τηρήθηκαν οι κανόνες όπως έπρεπε. Και γιατί να μην κάνουμε και μια επιτροπή έρευνας. Πιστεύω ότι όχι μόνο πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα, αλλά να εξεταστούν και οι δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν αυτά τα 7 τελευταία χρόνια. So, vielen Dank an die Kommission, Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή αλλά και του συναδέλφου για τη μεγάλη πειθαρχία που επέδειξαν στη συνεδρίαση. Ήταν πολύ σημαντικά όσα συζητήσαμε και νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε από εδώ και μπρο πώ θα χειριστούμε το θέμα. Πρόκειται για ένα ζήτημα πολύ σημαντικό που θίγει, ε, αφορά 400-500 χιλιάδες τουλάχιστον κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν αληθινά τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση, αυτό είναι βέβαιο. Έχουμε να κάνουμε με θέματα δημόσια υγεία, βασικά ζητήματα. Ιατρικά παρασκευάσματα τέτοιου τύπου δεν πρέπει να φτάνουν μέχρι την αγορά. Δεν πρέπει να βρίσκουν δηλαδή παραθυράκια τα οποία του επιτρέπουν να διατίθενται στον καταναλωτή, στον ασθενή και πρέπει να του ε, παρακολουθούμε πάντα, να κλείνουμε τα παραθυράκια αυτά και να επιβάλλουμε και τι σχετικές κυρώσει όποτε χρειάζεται. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη που αφορά τον απολογισμό τη αντιπροσωπεία τη επιτροπή μα στην Τουρκία. Το λόγο θα λάβει ο Γιολάινεν, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, στην επίσκεψη που έλαβε χώρα από τις 2 μέχρι 4 Νοεμβρίου το 2011 και παρακαλώ τώρα το Γιολάινεν να ε, λάβει το λόγο αφού πρώτα όμως αποχωρήσουν όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Ξέρω ότι είμαι πολύ φιλόδοξος, αλλά ξέρω ότι περιμένουμε και επισκέψεις και γι' αυτό θέλω να είμαστε στην ώρα μας έτοιμοι για να υποδεχθούμε την ε, επισκεπτρία μας. Ο Γιώλα έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επισκεφθήκαμε την Τουρκία διότι το κεφάλαιο που αφορά το περιβάλλον ε, ουσιαστικά είναι πάντα το ίδιο σε πραγματεύσεις για την ένταξη Παραμένει το ίδιο δηλαδή σε διαπραγματεύσει για την ένταξη του κράτου αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας υποδέχθηκαν με πολύ μεγάλη ε, φιλοξενία, είχαμε πολύ καλή υποδοχή, παρουσία απολών ε, από τους συνομιλητές μας, τα μέλη σχεδόν ολόκληρης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Επιτροπής Γεωργίας, μεγαλειώδης υποδοχή. Θεωρήθηκε δηλαδή πολύ σπουδαία υπόθεση η επίσκεψή μας ε, για τους Τούρκους ε, οικοδεσπότες μας. Έχει τεράστια ανάπτυξη η Τουρκία, 8-9% από ό,τι φαίνεται για δεύτερη χρονιά. Και υπάρχει βέβαια μοιραία η σύγκρουση, η ασυμβατότητα με τα θέματα του περιβάλλοντος. Ένα ζήτημα σημαντικό είναι αυτό της προμήθειας σε ενέργεια. Το έχουμε συζητήσει. Ενδιαφέρον είναι ότι η Ένωση Βιομηχάνων της Τουρκίας είναι εκείνη η οποία περισσότερο πιέζει για αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργεια και τι ανανεώσιμε πηγέ, από ό,τι ακόμα και η κυβέρνηση θα έλεγα. Η Τουρκία έχει διάφορες μορφές ενέργειας διάθεσή τη, ε, υδροηλεκτρικά, χρήση του, του άνθρακα, κάρβουνο δηλαδή. Σκοπεύει τώρα να σκευάσει και πυρηνικά εργοστάσια. Εμεί λοιπόν επισημάναμε ιδιαίτερα το μέλημά μα για την αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργεια και κυρίω τη στροφή προ τι ανανεώσιμε πηγέ. Ε, συζητήσαμε με τι περιβαλλοντικέ οργανώσει ε, την επαλήθευση τη συμβατότητα με το περιβάλλον που ε, ναι μεν προβλέπεται σε μια νομοθεσία, σε ένα νόμο τη Τουρκία, ο οποίο υπάρχει ισχύ αλλά δεν λειτουργεί, δεν εφαρμόζεται ουσιαστικά ή πάντω πολύ περιορισμένα και πρέπει ουσιαστικά να βελτιωθεί η υλοποίησή του. Συζητήσαμε επίσης ε, με το Υπουργείο Γεωργίας σε μια μεγάλη συζήτηση θέματα υγειονομικά, φυτοϊγιεινής, έχουν ε, αντιμετωπιστεί πολλά προβλήματα, λίγες είναι οι δυσκολίες όσο με το βορδινό κρέας της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Η Τουρκία όμως θα πρέπει να βελτιώσει ποντικά την σήμανση, την επισήμανση των προϊόντων, γιατί εκεί υπάρχουν προβλήματα. Για τη δημόσια υγεία συζητήσαμε ιδιαίτερα τα προϊόντα καπνού και το αλκοόλ, το ενοπνευματόδη, αλλά και τη ρήπανση, την ατμοσφαιρική ρήπανση στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως επίσης όμως ιδιαίτερα το κάπνισμα στο χώρο εργασίας αλλά και ε, στο κατοίκον, εν πάση περιπτώσει, στο εσωτερικό της κατοικίας του καθενός. Η Τουρκία δείχνει μεγάλη φιλοδοξία στην ε, διαδικασία αυτή των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μπαΐς, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο οποίος πάντοτε ήταν έτσι πολύ ε, πληθωρικός στην ε, στάση του, μας έλεγε πόσο σημαντικές ε, είναι οι αλλαγές που έχει φέρει η κυβέρνησή του στην ε, στάση της Τουρκίας ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ξέρουμε ότι και μας είπε ότι έχει μειωθεί η αποδοχή από, το, την κοινή γνώμη μέχρι και 35% τώρα από το 85% για την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε καμιά κάποια προσοχή και από πλευράς μας ως προς τη στάση μας προς την Τουρκία και τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Επίσης η ε, κυρία Ελένη Θεοχάρους από την Κύπρο σε μια συνεδρίαση Ε, είδε ότι στο τραπέζι της ήταν ε, μία ταμπελίτσα η οποία έλεγε ε, εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής διοίκησης. Βέβαια φαίνεται ότι αυτό ήταν απλώς μια δοκιμασία για να δούνε τις αντοχές της. Βγήκε εμπάσως η ίδια έξω σε ένδειξη διαμαρτυρίας και δεν αντιμετωπίστηκε το ίδιο φαινόμενο πλέον. Άρα φανταζόμαστε ότι στο δεύτερο ήμιση του έτους που θα έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουμε πάλι τέτοιου είδους τεστ αντοχής για το πώς θα χειριστεί πώς θα συμπεριφερθούν ε, οι Τούρκοι, πώς θα συμπεριφερθεί η Τουρκία στο θέμα της ε, Κύπρου. Πάση η περιπτώσει η Τουρκία είναι ένα σημαντικό κράτος, ένα μεγάλο κράτος. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα θέματα του περιβάλλοντος και περιμένουμε ότι θα προεράσει γρήγορα στην ενσωμάτωση όλη τη κύρια νομοθεσία για το περιβάλλον που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λάιρον. Ο κύριο Σκυλακάκη έχει το λόγο. Thank you, Mr. President. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη αυτή στην Τουρκία. Εγώ έθεσα διάφορα ιδιαίτερα ζητήματα. Είναι αλήθεια ότι η Τουρκία εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Και είναι επίση αλήθεια ότι πρόκειται για μια μεγάλη βιομηχανική δύναμη στην περιοχή μας. Από ό,τι φαίνεται, τα επόμενα 5 ή 7 χρόνια θα φτάσει στον ευρωπαϊκό μεσόρο όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι η Τουρκία δεν συμμετέχει και δεν έχει καμία ειδική πολιτική όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό το καταλάβαμε όλοι, γιατί εγώ το ρώτησα επανειλημμένος. Αυτό σημαίνει, συνεπώς, για την Νότια Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιταλία και ίσως και άλλες μεσογειακές χώρες Υπάρχει ιδιαίτερο κίνδυνο για διαρροή διοξιδίου του άνθρακα, γιατί όπω σα είπα, πρόκειται για μια μεγάλη βιομηχανική δύναμη, η οποία πολύ σύντομα θα βρεθεί στο δικό μα επίπεδο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και δεν έχει καμία σχετική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει απολύτω τίποτα για το θέμα, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ μετά από τι ερωτήσει που του έχω θέσει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Είναι σημαντικό γιατί έχει να κάνει με την ενέργεια, μπορεί να εξάγει ενέργεια η Τουρκία χωρίς να πληρώνει τίποτα για τις εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα και είναι και σημαντικό εξαιτία διαφόρων ειδικών προϊόντων τα οποία γεωγραφικά είναι εύκολο να εξάγει στους γειτονές της δηλαδή και τα οποία δεν λαμβάνονται οι υπόψεις στο benchmarking γιατί το σύστημα ανταλλαγών δεν έχει γεωγραφική πτυχή. Το benchmarking δεν έχει καμία γεωγραφική πτυχή. Είναι ένα τμήμα της Ευρώπης το οποίο είναι πλήρως προστατευμένο γεωγραφικά και ένα τμήμα της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Επειδή το τμήμα αυτό είναι πολύ κοντά στη χώρα μου, εμείς είμαστε δίπλα στην Τουρκία, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Υπάρχει και η Βουλγαρία που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, η Ρουμανία και άλλες μεζογειακές χώρες. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πολύ. Η κυρία Πλάμτορ έχει το λόγο. Παρακαλώ πάρα πολύ στο μάμος. Ευχαριστώ. Και εγώ συμμετείχα στην ε, επίσκεψη αυτή στην Τουρκία. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εδώ δεν θέλω να επαναλάβω τόσο επανή Πρέπει να σας πω ότι η Τουρκία βρίσκεται σε πλήρη οικονομική εξέλιξη και έχει επιπτώσεις πάνω στο περιβάλλον. Πρέπει να ζητήσουμε από τη χώρα αυτή συνεπώς να πάρει μέτρα έτσι ώστε να έχει μια πολιτική αντιμετώπιση των εκπομπών της διοξιδίου του άνθρακα για να μπορέσει έτσι να σεβαστεί και όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά το περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη και τη διαβούλευση με τους πολίτες, γιατί εμεί συναντηθήκαμε με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το περιβάλλον, συναντηθήκαμε και με επιχειρηματίες, Όλοι πρέπει να συμμετάσχουν σε μια διαβούλευση. Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να εκφραστούν όταν πρόκειται για άδειες όσον αφορά το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μια ακόμη παρέμβαση. Κυρία Γκίρλινγκ, παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ. Σύμφωνο με τον ε, Προεδρό μας, έτσι όπως ε, παρουσίασε τις ε, επαφές μας με την κυβέρνηση και με άλλους Όντω όπω ακούσατε, βρεθήκαμε και με επιχειρηματίε. Όμω θέλω να υπογραμμίσω κάτι που ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικό. Και αυτό ήταν ακριβώ οι επαφέ μα με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Πολύ σημαντικό αυτό για μα. Όταν πηγαίνουμε σε αντιπροσωπείε, ξοδεύουμε χρήματα, έτσι. Πάμε ένα σωρό από μας. Γιατί πάμε. Πάμε για να συναντηθούμε με ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται εκεί και δεν μπορούν να βρίσκονται εδώ. Αυτή την ευκαιρία όμως δεν τη χρησιμοποίησαμε. Με μία μη κυβερνητική οργάνωση συναντηθήκαμε στο τέλος του ταξιδιού μας. Θα ήταν μία ομάδα, αλλά τελικά ήταν μία περίπτωση μόνο. Και θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι ως Επιτροπή Περιβάλλοντος, όταν πηγαίνουμε σε αντιπροσωπείες, πρέπει να συναντιόμαστε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ίσως πρέπει να το φροντίζουμε από πριν να οργανώνουμε τέτοιες επαφές για να γίνονται. Γιατί αλλιώς δεν κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε και σίγουρα δεν παίρνουμε τις απαντήσεις. Αυτή τη φορά βρεθήκαμε μία κυβερνητική οργάνωση και στο τέλος του ταξιδιού. Θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει πολύ νωρίτερα στο ταξίδι μας. Άλλοι δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Χόσλιχαρτ και μετά επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να επαληθεύσουμε τα όσα λέει η κυβέρνηση με συγκεκριμένα παραδείγματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έχουμε δει όλα μας, τα έχουν γράψει, τα έχουμε διαβάσει, αλλά δεν επαληθεύεται τίποτε. Δεν βλέπουμε ένα αντικείμενο, δεν βλέπουμε τίποτε το απτό το συγκεκριμένο και αυτό είναι το πρόβλημα για μένα πάνω απ' όλα. Κύριος Λάινεν, δύο φράσεις μόνο πρόεδρε μια επίσκεψη στην Τουρκία είναι πάντα επίσκεψη στην Άγκυρα που εδρεύει η κυβέρνηση και στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που πράγματι λειτουργεί η κοινωνία. Και μέσα σε μια-δυο μέρε, όπω καταλαβαίνετε, το, πρόβλημα, το πρόγραμμα καθίσατε πολύ δύσκολο να τηρηθεί. Ε, Επίση, μη κυβερνητικέ οργανώσει στην Τουρκία δεν είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένε όπω στι δικέ μα χώρε. Υπάρχουν βέβαια μη κυβερνητικέ οργανώσει, αλλά όχι τόσο πολλέ. Δεν μπορούσαμε να δούμε πολλές επιμέρους μικρότερες οργανώσεις, μόνο τη γενική την ε, οργάνωση ομπρέλα που εκπροσωπεί τις ε, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Σε μια επόμενη επίσκεψη να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Ήταν πολύ δεξοδική, πολύ καλή εμπειρία που συλλέξατε. έτσι ώστε να μπορούμε και να αντιδράσουμε, να ζητήσουμε να αλλάξουν κάποια πράγματα και να περιμένουμε σε προσεχείς επισκέψεις ε, της αλλαγές, αλλά και σε άλλα κράτη βέβαια αντίστοιχα. Και θα ήθελα ε, τώρα να σταματήσω το θέμα αυτό για να καλωσορίσω την ε, Υπουργό για Τρόφιμα, Γεωργία και Αλληλεία της Δανίας, κυρία Μέντε Γκέρσκοφ, η οποία έχει έρθει για να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της Δανίας για την Προεδρία φιλόδοξο πρόγραμμα. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα επίσκεψη την πρώην συνάδελφο Τόριν Σμιτ, την Πρωθυπουργό της Δανίας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και διεξοδική παρουσίαση των θεμάτων, πολύ καλά προετοιμασμένη η Πρωθυπουργό και γι' αυτό σας καλωσορίσουμε και εσάς και πάλι εδώ έχουμε πολλά κοινά θέματα, έχουμε πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντο και εμεί ε, στην δική μα την ημερήσια διάταξη ε, ιδιαίτερα τι μας ενδιαφέρει η ε, αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας, η βιοπικιλότητα, η ηλεκτρονική επισήμανση, κρέατος και άλλων προϊόντων. Και βέβαια εδώ θέλουμε να συνεργαστούμε με το Ε, με το Συμβούλιο βέβαια για να προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε μια νέα Προεδρία, αλλά και εσείς είσαστε νέος Πρόεδρος, από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αλληλοβοηθούμε τους επόμενους έξι μήνες της Προεδρίας μας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και που μπορώ να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Προεδρίας μας. Έχουμε δουλέψει πολύ για την Προεδρία αυτή και καλό θα ήταν ευθύ εξ αρχής να σας τονίσω ότι αντιλαμβανόμαστε πως οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που μας περιμένουν είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Συνεπώς, πρέπει να αλληλοϊποστηριζόμαστε και να έχουμε ανοιχτή γραμμή για συνεργασία ανα πάσα στιγμή μεταξύ μας. Θα σας κάνω μια μικρή εισαγωγή για τις κύριες προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Εμείς θέλουμε να είμαστε μια υπεύθυνη, δυναμική, πράσινη και ασφαλής Ευρώπη. Γι' αυτό θα δουλέψουμε. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας και θέλουμε ένα μέλλον το οποίο οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά να είναι ασφαλές. Μετά την παρουσίαση του προγράμματος θα επεκταθώ λίγο περισσότερο όσον αφορά τα διάφορα θέματα που έχουμε στην ατζέντα μπροστά μας. Θα ετοιμάσουμε μία ατζέντα υπέρ της αηφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Θέλουμε ανάπτυξη και απασχόληση και εξαγωγές χωρίς να αυξήσουμε την κατανάλωση πόρων και ενέργειας. Και αυτό είναι εφικτό. Θέλουμε να προωθήσουμε την πράσινη ατζέντα. Αυτή είναι μια αναγκαία πρόκληση. Η πράσινη ανάπτυξη είναι αναγκαία για τη μελλοντική μας ευημερία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αλλά φυσικά πρέπει να επικεντρωθούμε επίσης και σε λύσεις που θα έχουν χαμηλό κόστος και που θα λαμβάνουν υπόψη την ανταγωνιστικότητα των εμπορικών μας επιχειρήσεων. Θέλουμε να επικεντρωθούμε λοιπόν στην πράσινη ανάπτυξη, κάτι το οποίο θα προσφέρει ευκαιρίε. Είμαστε σίγουροι. Χρειαζόμαστε ένα ελαστικό πλαίσιο για την πράσινη ανάπτυξη, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε καινοτομία και θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει και να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην τεχνολογία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει το δρόμο. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αδράξει την ευκαιρία αυτή της πράσινης ανάπτυξης, τότε το ρόλο αυτό θα τον αναλάβει κάποιος άλλος. Από τον Οκτώβριο που μας πέρασε, έχουμε τη συζήτηση και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής γίνεται και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της αναδιαμόρφωσης της κοινή γεωργικής πολιτικής, ώστε να ανταποκρίνεται στις ε, νέες ανάγκες, στις νέες προτεραιότητες και στις νέες προσδοκίες των Ευρωπαίων αγροτών, πολιτών, ε, καταναλωτών και φορολογούμενων. Είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε και αυτό. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ νωρί βέβαια για να μπούμε στις λεπτομέρειες όσον αφορά τα διάφορα στοιχεία κλειδί της μεταρρύθμισης, αλλά θα αναφερθώ μόνο στην απλοποίηση, το πρασίνισμα και τη συνοχή τη πολιτική μα κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα κάνει τη διαφορά. Επίσης, έχουμε και ένα άλλο στοιχείο προτεραιότητα και αυτό είναι η κοινή αλληλευτική πολιτική. Εκεί δοκιμάζεται η αντίληψή μας για την ε, πράσινη ανάπτυξη. Εδώ είναι που η οικονομία μας εξαρτάται πολύ περισσότερο από το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η ηγετική θέση όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και να ξεχρονίζουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι καταναλωτές μας πρέπει να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ότι τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι υγιεινά, υψηλής ποιότητας, ασφαλή και ε, προστατεύουν τα ζώα. Πρέπει να υποφεληθούμε από κάθε ευκαιρία που μας δίνεται για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια τροφίμων. Ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη προτεραιότητα ε, κατά την Προεδρία μας. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσουμε και τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση ε, όπως επίσης θέλουμε να δώσουμε μεγάλη σημασία και στην ασφάλεια των εισαγόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τροφίμων. Θα αναφερθώ τώρα σε συγκεκριμένες προτάσεις που ξέρω ότι εσείς εξετάζετε εδώ στην Επιτροπή σας. Όσον αφορά την πρόταση για τα τρόφιμα για βρέφη, και για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Εδώ θέλουμε να απλοποιήσουμε την τρέχουσα νομοθεσία που ισχύει από το 1989. Το Συμβούλιο λοιπόν δέχεται να εγκαταλείψει την έννοια των διατητικών τροφίμων όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη όμως έχουν κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά τον περιορισμό του εύρους εφαρμογής για τα τρόφιμα αυτά. Πιστεύει τα κράτη-μέλη ότι υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις και ότι χρειάζεται η ίδια νομική μεταχείριση για τα διατητικά τρόφιμα όπως και για εκείνα ε, όπως είχαμε μέχρι τώρα. Έχει ήδη γίνει συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δείχνει ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί. Τώρα όσον αφορά την Προεδρία μας, έχουμε σοβαρού λόγους να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λύση και συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Προεδρία ε, θα προσπαθήσει να πετύχει μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με τη συνεργασία βέβαια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Προεδρία ε, θέλει να συνεχίσει την καρποφόρα συνεργασία που έχει με τον εισηγητή και με την Επιτροπή σας γενικότερα. Επιτρέψτε μου τώρα, σύντομα, να υπογραμμίσω ποιες είναι οι απόψεις της Προεδρίας όσον αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ε, βοηδών και την ε, διαγραφή της ε, διάταξης όσον αφορά την σεθελοντική βάση σήμανση των βοηδών. Θα φροντίσουμε να υπάρχει πρόοδος και συμφωνία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Τώρα έχουμε κάτι άλλο. Την ευημερία των ζώων, την προστασία των ζώων. Είναι αποφασιστικής ε, σημασία και θα είναι στην ατζέντα της Προεδρίας. Στι 10 Νοεμβρίου του 2011 ο Επίτροπος Νταλή υπέβαλε έκθεση όσον αφορά την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Η Επιτροπή η έκθεση μάλλον αυτή της Επιτροπής ε, παρουσιάζει την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την εφαρμογή της ρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μεταφορά των ζώων και εντοπίζει ε, διάφορους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία ε, παρουσιάζονται. Η Προεδρία θα φροντίσει το Συμβούλιο να εξετάσει την έκθεση αυτή. Πρέπει επίσης να αντιληφθούμε ότι ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες έχουν υπογράψει στη σχετική ιστοσελίδα όσον αφορά τη, τον ανώτατο χρόνο μεταφοράς των ζώων. Αυτό βέβαια μπορεί να μην πρόκειται για νομική πρόταση, όμως είναι πολύ σημαντικό σινιάλο που μας στέλνουν οι καταναλωτές και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σε μας που νομοθετούμε. Επίσης, θα εξετάσουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την ευημερία των ζώων για την περίοδο 2012 με 2015, κάτι το οποίο έχει μόλις εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο στις συζητήσεις και έχει εγκρίνει την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του ε, του Μαΐου του 2010 σχετικά με την ε, αξιολόγηση του προγράμματος αυτού δράσης 2006-2010. Στα πλαίσια αυτά, η Προεδρία της Δανίας θα οργανώσει μια διάσκεψη με την Κομισιόν όσον αφορά την ευημερία των ζώων εδώ στις Βρυξέλλες, 29 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2012. Ιδιαίτερα για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, εφαρμογή και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ευημερία των ζώων. Εδώ θα συμμετέχουν ε, διάφοροι παράγοντες και αξιωματούχοι και εμπλεκόμενοι από την κοινωνία των πολιτών κλπ. Τώρα και κάτι που έχει να κάνει με την ε, ζωική παραγωγή και την ανθρώπινη υγεία. Εδώ ανταποκρινόμαστε στο πρόγραμμα δράσης για τις ε, νέες απειλές όσον αφορά την αντίσταση στους ε, μικροοργανισμούς. Εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι 25.000 άτομα στην Ευρώπη χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας αυτού του θέματος. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε. Και θα το κάνουμε αυτό όσο καλύτερα μπορούμε στον τομέα της υγείας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν έχουμε λάβει υπόψη μας τις δύο εκθέσεις που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Η διάσκεψη που έχει αυτό τον τίτλο «Καταπολέμηση της ε, αντίστασης των ε, μικροοργανισμών αυτών» θα λάβει χώρα στην Κοπεχάγη 14 και 15 Μαρτίου. Στόχος της διάσκεψης αυτής είναι να εξετάσει τις καλύτερες ε, πρακτικές για να αναπτύξουμε δράσεις κατά της αντίστασης αυτής. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια που είναι ένας πολύ βασικός ε, παράγοντας εξαγωγών, να παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση ενός συστήματος ε, εποπτείας του κρέατος. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ ελκυστικό να μιλάει κανείς για τον έλεγχο του κρέατος, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι Α, μπορεί οι ορισμένοι να το βρίσκουν ελκυστικό. Σεξι, λέει ο Μιλήτρια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των τροφίμων. Και βέβαια είναι και πολύ ακριβό για τους παραγωγούς μας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί. Και γι' αυτό και θα έχουμε μια διάσκεψη επίπεδου εμπειρογνωμόνων 2 και 3 Φεβρουαρίου για να συζητήσουμε ενδεχόμενες αλλαγέ στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Συνεπώς, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω διαβεβαιώνοντά σας για το ότι η Προεδρία της Δανία θα κάνει ό,τι μπορεί τους επόμενους μήνες προκειμένου να ε, προχωρήσει σε έναν καρποφόρο διάλογο μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων. Θα ολοκληρώσω αναφέροντας ένα πρόγραμμα της Δανίας, σίγουρα αναφέρθηκε σε αυτό ο Πρωθυπουργό μας, που ονομάζεται «Η Ευρώπη στη δουλειά». Νομίζω ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης, σαν αυτή μέσα στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να είμαστε αισιόδοξοι και να ξέρουμε ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση δουλεύοντας και ότι αυτό θα το κάνουμε με πράσινο τρόπο. Εγώ σας ε, διαβεβαιώνω ότι θα το φροντίσω αυτό και θα φροντίσω να θέσουμε στέρεα θεμέλια για την μελλοντική ευρωπαϊκή γεωργία, αλία και ασφάλεια τροφίμων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά θα ακούτε τα χειροκροτήματα. Σας ευχαριστούμε που παρουσιάσατε το φιλόδοξο πρόγραμμά σας, πολύπλευρο. Και αυτό που ιδιαίτερα σημείωσα εγώ και μου άρεσε, ε, κύριε Υπουργέ, είναι ε, το τελευταίο που είπατε για την Ευρώπη στη δουλειά. Την ε, Ευρώπη που δουλεύει. Γι' αυτό και βασίζουμε τις ελπίδες μας στη δικιά σας Προεδρία και ελπίζουμε ότι χάρη στην δικιά σας νομοθεσία, στις καλές προτάσεις που θα κάνετε, θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που υπάρχουν και έτσι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να εμπνεύσουν και πάλι με εμπιστοσύνη τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε και αυτό ακριβώς βλέπουμε στο πρόγραμμά σας. Οι συνάδελφοι πάντως έχουν ερωτήσεις να σας κάνουν. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ξεκινήσουμε συνεπώς ευθύ αμέσως. Τρία λεπτά προτείνω με δύο κύκλους ε, ερωτήσεων προκειμένου να μην μαζευτούν πολλέ. Λοιπόν, τρία λεπτά έχει ο καθένα για τις ερωτήσεις. Λίντα Μακάβεν πρώτα. Και μετά η Κρίστε Σάρδεμόσα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω δανέζικα. Ξεκινάει η κυρία Σάλτερ Μόζε, μια που έχουμε εδώ ε, τον εκπρόσωπο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ μαζί μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλες τα δανέζικα, κυρία Σάλτερ Μόζε. Και να ξέρετε ότι για μένα είναι δύσκολο να επιφέρω κριτική στο πρόγραμμα της Δανέζικης Προεδρίας, γιατί το βρίσκω πραγματικά φιλόδοξο. Και συμφωνώ με αυτό που λέει η Προεδρία, ότι δηλαδή η Ευρώπη πρέπει να ανασκουμποθεί και να μπει στη δουλειά. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω και κάποια κριτική. Και θέλω να ρωτήσω πώς πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη θα καθίσουν να δουλέψουν έτσι ώστε να φανεί ότι η Ευρώπη δουλεύει επίσης. Γιατί συχνά είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε μια καλή νομοθεσία, το πρόβλημα όμως είναι πώς θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η καλή νομοθεσία από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν ρωτάω στο Συμβούλιο πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα. Δεύτερη ερώτηση. Η αντίσταση αυτή στα αντιβιωτικά. Όλοι γνωρίζουμε εδώ στην Επιτροπή αυτό ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το θέμα αυτό για την ανθρώπινη υγεία. Τι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εσείς θα αναλάβετε στον τομέα αυτό. Ξέρω ότι εκφράζονται ανησυχίες, ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην Ευρώπη γι' αυτό. Οι ευρωπαϊκές χώρες ε, της Βόρειας Ευρώπης ίσως είναι πιο συντηρητικές σε σχέση με εκείνες της, βόρειας, της Νότιας Ευρώπης. Ρωτώ λοιπόν πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα. Έπειτα για τα τρόφιμα. Εδώ έχουμε υπογραμμίσει την διφενόλη α στα τρόφιμα, γιατί η ουσία αυτή, ναι, που είναι στις συσκευασίες, στις συσκευασίες των τροφίμων, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που περνάει δηλαδή η ουσία αυτή και στα τρόφιμα μερικές φορές. Ορισμένες χώρες προβλέπουν να απαγορεύσουν την ουσία αυτή εσείς στην πράξη πώ θα τα προχωρήσετε όλα αυτά. Πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμά σας και είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς στα πλαίσια των νομοθετικών προτάσεων που θα γίνουν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντελάγκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση στον τομέα των τροφίμων. Οπότε κατάλαβα, ε, προβλέπετε μια αναθεώρηση της ε, οδηγίας ε, για το τρόφιμα. Καταλάβα ότι είναι προτεραιότητα για τη δική σας προεδρία. Φυσικά δεν μπορώ να προβλέψω την ψηφοφορία που θα γίνει εδώ, αλλά ήδη μπορούμε να διαβλέψουμε με τη βάση των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί πώς, ποια είναι τα επίμαχα ζητήματα. Εγώ θα ήθελα να τονίσω δύο που θα ήθελα να μας ενημερώσετε για το ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση ε, στο Συμβούλιο. Το ένα είναι το, οι δίαιτες ε, πολύ λίγων θερμίδων. Η πρόταση της Κομισιόν είναι να αποκλειστούν όλα τα προϊόντα χαμηλών ε, θερμίδων από την νομοθεσία αυτή και να τοποθετηθούν στην γενική νομοθεσία. Εάν δούμε όμως τις τροπολογίες που έχει υποβάλει η Επιτροπή μας, εμάς μας ανησυχούν πολύ τα προϊόντα πολύ χαμηλίων θερμίδων. Δηλαδή είναι μόνο 400 με 800 θερμίδες ημερησίως. Κατά κάποιο τρόπο θέλουμε εμείς να μείνουν στο ειδικευμένο πλαίσιο. Ε, τι που βρίσκεται η κατάσταση στο Συμβούλιο και δεύτερο είναι τα γάλα ανάπτυξη στον τομέα των βρεφικών τροφίμων. Οπότε κατάλαβα η Δανία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου αυτά τα προϊόντα δεν κυκλοφορούν στην αγορά γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει ζήτηση για αυτά. Αλλά έχουμε τα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη όπου κυκλοφορούν αυτά τα προϊόντα. Προσωπική μου γνώμη είναι πως τα προϊόντα αυτά για τα παιδιά πάνω από την, ε, την ηλικία του ενό έτου μπορούν να παχθούν στην γενική νομοθεσία και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία. Αλλά η Κομισιόν δεν μου απαντά ε, για το τι θα συμβεί αν η οδηγία αυτή απορριφθεί και άρα αυτά τα προϊόντα τοποθετηθούν στην αγορά υπό την ε, οριζόντια οδηγία. Θα αποκλειστούν δηλαδή όλα αυτά τα προϊόντα ή θα μπουν στην αγορά υπό αδιαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. Πού βρίσκεται λοιπόν η πρόοδος στο Συμβούλιο. Και αν μπορούσατε να μας ενημερώσετε για όλα τα άλλα θέματα σε σχέση με την Πάρνετ που σας απασχολούν, όπως η γλουτένη ίσως, θα ήταν καλό λοιπόν για αυτό να έχουμε μια γενική εικόνα. Και νομίζετε πως θα καταφέρετε να φτάσετε σε, σε συμφωνία υπό τη δική σας Προεδρία. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Η Φρεντερή Κρίστα κάνει την πρώτη ερώτηση για μας. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσκοφ με το πολύ δύσκολο όνομα. Ε, πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Αυτό δεν έχει σχέση με το σημερινό θέμα, αλλά μιλούσαμε χθε με εκπροσώπους ε, των ε, γυναικών στην, στο Προεδρία μας, αλλά η Δανία τα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι άλλοι. Είδαμε την Πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα, την Υπουργό Γεωργίας τώρα, την Υπουργό Υγεία το απόγευμα σήμερα. Νομίζω ότι για την ώρα οι αντιπροσωπεύονται πολύ καλά στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ για τις προτεραιότητες που μας ε, ε, περιγράψατε εδώ. Ήταν βέβαια μια πρώτη εικόνα, αλλά ε, θέλησα και διάβασα το έγγραφο της Προεδρίας για την πράσινη οικονομία, την ανταγωνιστικότητα. Το είπατε με αυτό το μήνυμα του σλόγγαν ε, που αναφέρθηκε η Ευρώπη στη δουλειά. Ε, το status quo δεν είναι πλέον υποφερτό, το διαπιστώνουμε καθημερινά. Μετά από την παρέμβαση της κυρίας Δελάνγκη για την πρόταση για την οποία είμαι εισηγήτρια, μπάρν και συγκεκριμένα τρόφιμα, μου επιτρέπει να επανέλθω σε αυτό το θέμα, ότι να σας πω ότι έχουν κατατεθεί 500 τροπολογίες στις τρεις ε, ε, επιτροπές που είναι αρμόδιες, για να σας ε, εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι το θέμα και πόσο ζωντανό, πόσο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει και θα ήθελα να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει στο Συμβούλιο και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε για όλα αυτά τα επίμαχα και προβληματικά θέματα όπως ε, οι δίαιτες ε, ε, με πολύ λίγες θερμίδες ή τα βρεφικό γάλα. Τώρα ένα από τα άλλα σας σλόγγαν για τη Γεωργία είναι η Ευρώπη η εξαγωγική. Δεν νομίζετε πως θα έπρεπε επίσης να εξασφαλίσουμε τα μετόπιστα, δηλαδή να φτάσουμε σε κάποιο είδος αυτή επάρκειας. Εγώ είμαι φιλελεύθερη και δεν δουλεύουμε με παπαγορεύσεις, αλλά βρίσκω παράξενο να βλέπω όλα αυτά τα προϊόντα, όλα αυτά τα φρούτα, ε, λαχανικά στα σούπερ μάρκετ μας που έρχονται από τις τέσσερις γωνιές του ορίζοντα ε, και για το περιβάλλον είναι πολύ επιβλαβές αυτό, επιβαρυντικό. Και έπειτα μετά από την ψηφοφορία που κάναμε στο Στρασβούργο θα κάνετε κάτι ώστε να περιορίσουμε την ε, τροφική σπατάλη για τα τρόφιμα τα οποία είναι αναλώσιμα και έχει αποτελέσει αυτό πρωτοσέλιδο τίτλο στην, στο Βέλγιο με την έκθεση Κορώνα 80 ε, εκατομμύρια τόνοι σπατάλης ετησίως και είναι ένα νούμερο που θα διπλασιαστεί όπως προβλέπετε με το 2020 και αυτό είναι φυσικό και ανυπόφορο. Θα ήθελα λοιπόν να, κάνει, να λάβει κάποια πρωτοβουλία και Τέλος, για να ολοκληρώσω, αναφέρεται στο έγγραφό σας τον πολύ σημαντικό ρόλο της επιστηστικής ε, ε, τη βοήθεια και των τροφίμων με τα μέτρα που προτείνετε, τι έχετε υπόψη σας, τι θέλετε να κάνετε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι το βασικό τερό κομμάτι, είναι ανάμεσα στο 80 και 90% στην Ευρώπη και είναι πολύ συχνά δύσκολα τα πράγματα. Τι σημαίνει ισχυρισμός ε, τροφή, ε, διατροφής για την ΕΦΣΑ. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Ε, γι' αυτό και οι δράσεις μας θα πρέπει να είναι οριζόντιες για τις μικρομεσαίες. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρίση. Ισά του Χάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ την Υπουργό που ήρθε να συζητήσει. Θέλω να κάνω μια ερώτηση για την περιπολιτική πτυχή της γεωργικής πολιτικής που είναι ο ευτροφισμός ορισμένων θαλασσίων περιοχών όπως η Βαλτική θάλασσα και οι ακτές της που έχουν το πρόβλημα του ευτροφισμού λόγω των διαρροών διαφόρων τροφικών ουσιών της Γεωργίας. Η πολύ κακή κατάσταση της θάλασσας αυτής οφείλεται ότι ο βυθός δεν έχει πια οξυγόνο λόγω του ευτροφισμού είναι το, η μεγαλύτερη θάλασσα στον κόσμο ανεφοξυγόνου στο βυθό. Και η γεωργία είναι η, βασικός, η βασική πηγή ε, ουσιών ευτροφισμού στην Βαλτική θάλασσα και όχι μόνο. Είναι μια παραμελημένη, ξεχασμένη πτυχή της ε, ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε για την βελτίωση της οικολογικής κατάστασης της Βαλτικής θάλασσας και των πολλών ποταμών χωρίς μια νέα προσέγγιση στη γεωργική πολιτική. Και επειδή η Βαλτική θάλασσα είναι πολύ ε, γνωστή και για τους Δανούς, και προσφυλής και στους Δανούς, θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτή είναι μια πτυχή για τη Δανική Προεδρία ή όχι όταν ε, θα ασχοληθείτε με την ε, μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστούμε κυρία Χάση. Κρίστα Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ την Υπουργό που ήρθε σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία βεβαίως ιδιαίτερα μεριμνά για το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη της γεωργικής ε, ε, του γεωργικού τομέα την αναφέρατε και εσείς, έχει ιδιαίτερη σημασία και για το περιβαλλον και για τη δημόσια υγεία φυσικά. Την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, την αναφέρατε μόνο ακροθυγώς και όχι σε λεπτομέρειες. Είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό για μένα να κοιτάξουμε με την μεταρρύθμιση αυτή το τι μπορούμε να προσφέρουμε και για τις μεγάλες επιφάνειες και για την διασταυρούμενη συμμόρφωση, την cross compliance. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να προσμετρήσουμε και να συμβάλλουμε στο να μπορούν τα κράτη-μέλη να ελέγχουν καλύτερα τη διασταυρούμενη συμμόρφωση και στο μέλλον και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό ισχύει και για την προστασία των ζώων, ιδιαίτερα δε για τη μεταφορά ζώων. Έχουμε πολλά ε, ηλεκτρονικά μηνύματα ε, ανθρώπων που μεριμνούν για την προστασία της ευημερίας των ζώων που διαμαρτύρονται για τι ε, μεταφορέ σε μεγάλε αποστάσει ζώων και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο έλεγχο και ιδιαίτερα ε, να ενισχυθεί ο έλεγχος στι συνθήκες μεταφορά ζώων προ το ε, σφαγείο. Πριν από χρόνια θεσπίστηκε η νομοθεσία σχετική με την φυτογενή, με τη φυτοπροστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι θα έχουμε το 2012 τη σχετική αναθεώρηση, κυρία Υπουργέ, και γι' αυτό παρακαλώ να φροντίσετε στο ε, επίπεδο του Συμβουλίου να προχωρήσουν αρκετά γρήγορα οι εθνικές διαδικασίες εφαρμογή, εισαγωγή ε, στο εθνικό δίκαιο για να ε, υλοποιηθεί πολύ γρήγορα αυτή η νομοθεσία. Και επίσης τελευταία παρατήρηση όταν παράγονται σε συστήματα κλοβών αυγά ε, που δεν ανταποκρίνονται, δεν τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ομοθεσίας, παρακαλώ με έτσι ώστε να μην μπαίνουν στην αγορά μας, να μην έρχονται στην αγορά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιούργισεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Γιώργινσεν. Και ευχαριστώ πολύ και την Υπουργό που ήρθε εδώ. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ στις Βρυξέλλες. Μπορώ να πω και στους συναδέλφους ότι γνωρίζω την Υπουργό πολύ καλά από τη Δανία ήδη καλύτερο σύμμαχο για τους επόμενους μήνες, για τη δουλειά μας και σε σχέση με το Συμβούλιο δεν το που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που είστε εδώ. Και πρώτος, πρώτη παρατήρηση, ερώτηση, σχόλιο που έχει να κάνει και με το προσθήνισμα της ε, ΚΑΠ, της κυρίας γεωργικής πολιτικής. Είπατε κι εσείς ότι δεν μπορείτε να μπείτε, να επισέλθετε σε πολλές λεπτομέρειες. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξή, μήπω θα μπορούσατε να μα πείτε δύο λόγια για τι ε, αρχέ, τι γενικέ αρχέ τι οποίε σκοπεύετε να εφαρμόσετε, γιατί είναι πολλέ οι οργανώσει ε, ε, που έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για το ότι ενδεχομένω να ξεπλύνουμε την ΚΑΠ με πράσινο χρώμα να πάρει έτσι μια ελαφριά πράσινη απόχρωση, αλλά ίσω να μην είναι ουσιαστικό το πρασινισμά τη. Ποιε είναι οι βασικέ αρχέ λοιπόν που θεωρείτε ότι χρειάζονται για να μπορέσουμε πράγματι να εξασφαλίσουμε το πρασίνισμα. Επίση, δε, ε, και ευχαριστώντα σα βεβαίω ε, για την ε, ευχαριστώ που αναφέρατε την εκστρατεία που είχα ξεκινήσει στο ίντερνετ. Έχουμε πάρα πολλέ τώρα υπογραφέ. Πολλοί είναι οι συνάδελφοι από την Επιτροπή μα που αγωνίστηκαν επίση ε, στην υπόθεση αυτή της, ε, του 8 Θα ήθελα να συμπληρώσω ακόμη ε, το πλωστάσιο των επιχειρηματών σας με κάτι ακόμη, ότι ο Επίτροπος Νταγή βέβαια δύσκολα δυσκολεύτηκε ή δίσταζε να δεχτεί τέτοιε προτάσει και να τι προβάλλει στο Συμβούλιο. αλλά οι δύο προηγούμενοι Κυπριανού και Βασιλείου ε, Επίτροποι είχαν υποσχεθεί, δεν είχαν πει να δούμε και βλέπουμε, όχι, είχαν υποσχεθεί ρητά να υποβάλουν πρόταση πριν από το τέλο τη προηγούμενη θητεία ακόμη και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμη και ο Μπαρόσο μάλιστα, ο οποίο ε, είναι ο ε, προϊστάμενο ουσιαστικά αυτών των δύο επιτρόπων ε, έχει πρόβλημα διότι δεν έχει ε, ε, εκτελεστεί, δεν έχει υλοποιηθεί η υπόσχεση που από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Chris Davis και ο κύριος Σλούιτσερ για να κλείσει ο κατάλογος των αγορητών. Κύριε Davis, Πρόεδρε, ξέρω βεβαίως ότι είναι τεράστιο το χαρτοφυλακιά σας, ε, κυρία Υπουργέ, και για τα θέματα της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, την γεωργική πολιτική και μεταρρυθμισή της που με ενδιαφέρει ιδιαίτερω, θα ήθελα να πω το εξή. Βλέπω ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική σε υπουργικό επίπεδο δεν λαμβάνει από ό,τι φαίνεται την ίδια ε, τον ίδιο βαθμό προτεραιότητας, δεν αντιμετωπίζεται με την ίδια δηλαδή ε, σπουδή όπως θα θέλαμε. Ενώ ταυτόχρονα όμως ε, κάνουμε πολύ μεγάλες ζημιές στις μας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει η αλληλευτική πολιτική να προχωρήσει σε μια βαθύτατη μεταρρύθμιση, μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Ερωτώ όμως, έχετε επαρκή πολιτική υποστήριξη, έχετε αρκετή υποστήριξη από τους Πρωθυπουργού της Ευρώπης για να προχωρήσει στις αλλαγές που χρειάζονται. Δεν θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να κάνει μια διακήρυξη αρχών, να προβεί σε μια διακήρυξη αρχών για τα θέματα αυτά, για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής, ώστε να είναι ξεκάθαρο και σε κάθε επίπεδο, σε κάθε στρώμα της κυβερνητικής διαστρωμάτωσης, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό της μεταρρυθμίσης ε, αλληλευτικής πολιτικής και ότι δεν είναι κάτι δευτερεύον που θα μπορούσαν να σπρώξουν κάτω από το χαρλί. Και πιστεύω ότι μέχρι τώρα στην κοινή αλληλευτική πολιτική το κύριο πρόβλημα ήταν η ετήσια συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας το Δεκέμβριο, που, όπου, κατά την οποία κατανέμονται ποσοστώσεις από τους υπουργού χωρίς καμία ουσιαστική μελέτη και ορθολογική ε, σκοπιά. Λυπούμε λοιπόν, αλλά διαπιστώνω δυστυχώς ότι είναι πολλοί υπουργοί στο Συμβούλιο με τους οποίους θα έχετε να κάνετε κατά τη θητεία σας εδώ που δεν θα είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν σε κάτι. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ιδέες κάποια σχόλια. Ευχαριστώ τον Κρις και τελευταίο ο κύριος Σλίτσαρ. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Επίσης λέει ο πρόεδρος. Και χαίρετε και πάλι, όπως θα φαντάζεστε, και εγώ θα μιλήσω για την ε, μεταφορά ζών των ζώων. Μιλήσαμε για το 1 εκατομμύριο υπογραφών. Η κυρία Κλάς ήδη εξέφρασε τις θέσεις μας, τα όρια. Υπόθηκε επίσης ότι έχουν δοθεί υποσχέσεις από τους επιτρόπους, αλλά περιμένουμε να δούμε και ουσιαστική εφαρμογή και εκτέλεση βέβαια των υπεσχημένων, αλλά και η υλοποίηση της νομοθεσίας, γιατί έχουμε διπλό πρόβλημα εδώ πέρα. Και το ότι δεν εισάγεται η νομοθεσία, αλλά και δεν εφαρμόζεται όταν υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Λοιπόν, να επικεντρωθούμε στην ε, ε, εφαρμογή της νομοθεσίας, μας λέτε πολλές φορές, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα, γιατί εάν δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία, το πιο απλό είναι να μειωθεί ο χρόνος μεταφοράς ή να υπάρχουν τόποι αναψυχή και ανάπαυση και να ε, αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα εφόσον δεν υλοποιείται σωστά η νομοθεσία. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι έχουμε υπογραφές, ένα εκατομμυρίο υπογραφές. <laughs> ως προς, την, ε, ως προς τα αντιβιωτικά, την αντίσταση στα αντιβιωτικά, Έχουμε πολλά προϊόντα τα οποία ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τρόπο διαφορετικό και θα ήθελα να μου πείτε για τα γενετικά τροποποιημένα για τα οποία έχουμε ένα εκατομμύριο υπογραφέ, τι στάση περιμένετε ότι θα τηρήσει το Συμβούλιο. Δημόσιε προμήθειε. πολλά θέματα μα απασχολούν εκεί και βεβαίω θα πρέπει να προαχθεί ως το δυνατόν η δυνατότητα συμμετοχή ε, στι αγορέ ε, κατά τρόπο ορθολογικό και των μικρότερων και τοπική εμβέλεια γεωργών. Εμεί έχουμε και πολλέ μάλιστα προσφυγές στα δικαστήρια στην πατρίδα μου, εκεί όπου προσπαθούν ε, οι δημοτικές αρχές ε, να διαφυλάξουν ή να διευκολύνουν την πρόσβαση των ε, τοπικής εμβέλειας παραγωγών στις συμβάσεις αυτές δημόσιων προμηθειών, αλλά εναντίον των οποίων γύρονται αγωγές και προσφυγές για λόγους διακριτικής μεταχείρισης. Αυτά λοιπόν όλα πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις σας. Πόσες ώρες έχουμε, Πρόεδρε, να προσπαθήσω να απαντήσω. Έχει, είναι πολύ σημαντικές οι ερωτήσεις σας και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τις απαντήσω. Πολλές ερωτήσεις αφορούσαν ε, την ευημερία των ζώων. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό εμείς ε, της Δανικής Προεδρίας να θέτουμε τις συζητήσεις ε, κατά τη διάρκεια της, της Προεδρίας. Ξεκινήσαμε συζήτηση για τις μεταφορές, για την δήλωση της Επιτροπής για την ευημερία που μπορεί να οδηγείται από άλλα πράγματα, δείκτες για την ευημερία των ζώων. Όλα αυτά ε, θα γίνουν και θα γίνει και διάσκεψη στην Κοπενχάγη για το θέμα αυτό. Ελπίζουμε πως θα έχουμε και συμπεράσματα του Συμβουλίου για αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό και μπορώ να σας πω επίσης πως ε, συνειδητοποιώ ότι κάποιοι κανονισμοί που έχουν γίνει στο παρελθόν τελικά φάνηκε ότι ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Γιατί ανέφερε η κυρία Κλάς για τις, ε, ο, ο, για οτόκες, ορνηθες που ανέφερε η κυρία Κλάς ε, είπαμε για να στέγαση. Πρέπει να κατασκευάσουν οι, οι πτυνοτρόφοι νέες συστοιχίες, νέους κλωβούς, και ούτω καθεξής. Όταν έχουμε λοιπόν μικρές ε, περιόδους εφαρμογή ε, σταματάει στη μέση το πρόγραμμα. Θα πρέπει γι' αυτό ε, να, να σκεφτούμε έναν διαφανή τρόπο εφαρμογής, έτσι ώστε τα κρατη να μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα τους θέσουμε για το πού έχουν φτάσει, πώς έχουν προχωρήσει. γιατί είναι τελείως απαράδεκτο ε, ορισμένες χώρες ε, να ε, να μην εφαρμόζουν τις οδηγίες και επίσης για τις οτόκες όρνηθες η Κομισιόν θα ξεκινήσει η διαδικασία κατά παράβαση κατά 14 κρατών μελών. Μα δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε αυτό, αλλά από την δική μου εμπειρία είναι πολύ γρήγορη δράση από την Κομισιόν αυτή. Και στην ε, συζήτηση ε, βλέπουμε ότι το θέμα είναι πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Τώρα, αν είναι διαφορετικό το σύστημα, ναι, είναι, υπάρχει τεράστια διαφορά όταν τα κράτη-μέλη ε, ελέγχουν ε, τα συστήματα. Εμείς ε, που θεωρούμε ως Προεδρία, είναι μια πρωτοβουλία περί ελέγχου που λέγεται One Health, αλλά συνειδητοποιούμε ότι αν έχουμε μια απόφαση για έλεγχο που θα καλύπτει πολύ περισσότερο έδαφος, θα έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε ενότητα σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό που σκεφτήκαμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχουμε για τα αντιβιωτικά. Πόσα ε, χρησιμοποιούνται, πώς χρησιμοποιούνται, γιατί υπάρχουν δύο διαστροματώσεις εδώ. καταρχήν, ποια είναι τα, ε, ποια, ποιες, ποιοι είναι οι όγκοι που χρησιμοποιούνται και ποιος είναι ο κίνδυνος στο συγκεκριμένο αντιβιωτικό να μετατραπεί σε κίνδυνο. Γιατί αυτό που χρειάζεται να δώσουμε στο μέλλον στους πολίτες μας είναι η δυνατότητα θεραπείας. Και θα ήταν φρικτό αν χρειαστεί να διώχνει το κόσμο στα ε, νοσοκομεία μόνο και μόνο επειδή έχουμε κάνει υπερβολική χρήση αντιβιωτικών στο παρελθόν. Ε, θα, θα εστιάσουμε την προσοχή μας πολύ στο θέμα των αντιβιωτικών κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Τώρα, είμαι πολύ αισιόδοξη και έχω μια συγκεκριμένη προσδοκία ότι θα γίνει πρώτη Θα υπάρξει συμφωνία πρώτης ανάγνωσης ε, σε αυτό το θέμα που είναι πρώτα στο πρωταρχικό του στάδιο, στο αρχικό του στάδιο και στο Συμβούλιο. Γνωρίζω πως υπάρχει μεγάλη στήριξη στο Συμβούλιο όταν πρόκειται για την πολυεθνική. για το VLCD. Αλλά πάντως είναι ακόμα υποσυζήτηση, δεν έχει τελειώσει τίποτα, δεν έχουμε καταλήξει. Και επίσης με ρωτήσατε για τη γλουτένη. Αυτό που είναι σημαντικό και είναι σημαντικό στο Συμβούλιο είναι η προστασία του κόσμου που πάσχει από δυσανεξία στη γλουτένη θα πρέπει να διατηρηθεί. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος που πάσχει από δυσανεξία στη γλουτένη να έχει το ίδιο επίπεδο προστασίας που έχει σήμερα. Ίσως αυτό να έχει να κάνει με την ε, ετικετοθεσία, τη σήμανση. Ε, θα δούμε αν θα το περιλάβουμε στο πεδίο εφαρμογής οδηγίε. αλλά θα δούμε πού θα καταλήξουμε για αυτό το θέμα. Τώρα, πώς θα κάνουμε τα κράτη-μέλη να δουλέψουν. Καταρχήν να σας πω ότι εντάξει, δουλεύουνε. Νομίζω πως δουλεύουνε και η Ευρώπη στη δουλειά σημαίνει πως όλοι δουλεύουμε. Ε, εντάξει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε οικονομική κρίση. Ωραία, δύσκολη καιρή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δουλεύουμε. Ε, νομίζω πως τα όσα είδαμε ως δανεική Προεδρία, εμείς διαρκώς συναντάμε κόσμο που πραγματικά θέλει να κάνει κάτι και να αλλάξει τα πράγματα και να προχωρήσει. Αλλά πιστεύω επίσης πως θα είναι σημαντικό, όπως ανέφερα, Ε, όπως για την προστασία των ζώων ας πούμε, στους κανονισμούς να υπάρχουν ε, ε, τρόποι να προχωρήσουμε με διάφορες στάσεις στο δρόμο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλη η Ευρώπη θα κινηθεί και θα προχωρήσει. Απόβλητα τρόφιμα, ναι. Συμφωνώ, είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Ξέρω και σας ευχαριστώ πολύ το Κοινοβούλιο που έθιξε αυτό το σημαντικό θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη στην Ολομέλεια από ό,τι κατάλαβα εδώ Δεν μπορώ να σας δώσω πολλές πληροφορίες για σχετικές ε, πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο για την ώρα. Ε, έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου από το Δεκέμβριο για αυτό το θέμα και μπορώ να σας πω από τη δανεική προοπτική ότι εμένα με ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Ας πούμε θα μπορούσε να μιλήσουμε για οργανικά τρόφιμα, για βιολογικά τρόφιμα. Βιολογική κουζίνα, μαγειρική, να επιμείνουμε γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι είμαστε τμήμα μιας παγκόσμια, ενός παγκόσμιου, μια παγκοσμιοποιημένη κοινότητας και μέσα σε μια τόσο δύσκολη οικονομική κρίση χρειαζόμαστε χρήματα που να έρθουν και εκτός Ευρώπης. Χρειαζόμαστε εξαγωγές και γι' αυτό είναι ένας τρόπος για να το πετύχουμε. Η κυρία Χάση ρώτησε για συστατικά ευτροφισμού στην ε, Βαλτική. Αλλά η Βαλτική είναι μία από τις πιο προβληματικές θάλασσες που έχουμε και γνωρίζουμε πως η γεωργία είναι μέρος της λύσης. Ήταν μέρος του προβλήματος και τώρα πρέπει να είναι μέρος της λύσης. αλλά πολλά νομίζω ότι ρυθμίζονται μέσω του οδηγία για το νερό Και όταν μιλάμε για την κοινή γεωρική πολιτική και τη μεταρρύθμιση τη, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν στοιχεία πρασινίσματο, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τα διάφορα συστατικά. Και την ερώτηση του κύριου Γιώργης για το πρασίνισμα. Ε, είναι πολύ σημαντικό το να εξασφαλίσουμε ε, ότι θα υπάρχουν αποτελέσματα μέσω αυτού του πρασινίσματος, να τα δούμε όλα τα αποτελέσματα. Όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή η, από τις επιδοτήσεις στον πρώτο πυλώνα μόνο το 70% πρέπει να καταβληθεί και το υπόλοιπο 30% πρέπει να πρασινίσει. Πρέπει να πρασινίσεις για να πάρεις και το υπόλοιπο 30% και υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που ε, βελτιώνουν και δίνουν ε, κίνητρα για να πρασινίσει ακόμη περισσότερο. Θα το συζητάμε στο Συμβούλιο για την διαφοροποίηση της, ε, των καλλιεργιών, των, της ποράς. Αλλά Ίσως χρειάζεται να έχουμε περισσότερα σε αυτό το, την δυνατότητα επιλογής, να είναι πιο συγκεκριμένο το ποια χώρα κάνετε. Όταν μιλάμε για πρασίνισμα, σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουμε διαφορετικά εδάφη, διαφορετικό κλίμα, διαφορετικές καταστάσεις που μπορεί να απαιτούν διαφορετικές απαντήσεις. Μια άλλη απάντηση θα μπορούσε να είναι να δούμε το δεύτερο πυλώνα, να δούμε πόσο πρασίνισμα χωράει εκεί. Δεν μπορώ να σας δώσω όμως εγώ συμπεράσματα γιατί αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει ακόμα στο Συμβούλιο. Είναι απλά κάποιες ιδέες που προσπαθώ να καλύψω. Για τον κύριο Ντέιβις, για την μεταρρύθμιση της αλίας. Ρωτήσατε να υπάρχει πολιτικό ενδιαφέρον. Αν δείτε την πρόταση της Κομισιόν, θα δείτε την πιο βιώσιμη μεταρρύθμιση της αλίας που εγώ τουλάχιστον έχω δει. Βιωσιμότητα είναι θεμελιώδης αξία που διαπερνά ολόκληρη τη μεταρρύθμιση. Πρέπει να καλυφθούν βέβαια ζητήματα στον τομέα τη αλίας, αλλά έχουμε προχωρήσει πολύ στις συζητήσει που έχουν γίνει μέχρι στιγμή. και νομίζω πως εάν ήσασταν κάπω αρνητικός για τις συζητήσει στο Συμβούλιο όταν, μιλά... Ε, ε, όταν μιλήσαμε για τα ΤΑΚ, Έγινε ωστόσο συζήτηση το Δεκέμβριο και για το κατά πόσο θα πρέπει να ανασταλεί το πρόγραμμα διαχείρισης για τη Βόρεια Θάλασσα και εσείς με ρωτήσατε τι γίνεται στο Συμβούλιο. Δεν το ανέστειλε το Συμβούλιο το πρόγραμμα διαχείρισης. Διατήρησε το στόχο βιωσιμότητα στη Βόρεια Θάλασσα χωρίς να γίνει καμιά συζήτηση ακόμα για τα ψάρια στη δική μας Προεδρία. Θα γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα. Θα έλεγα ότι υπάρχει πολιτικό ενδιαφέρον. νομίζω πως ε, κατανάλωσα πολύ χρόνο, αλλά υπήρχαν πολλά ζητήματα σημαντικά για τα οποία ήθελα να μιλήσω. Βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε και αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που είναι τόσο σημαντικά. Είναι δύσκολες οι εποχές και δύσκολα τα προβλήματα. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Κύριε να έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως να επαναλαμβάνονται κάποιες ερωτήσεις. Πάντως εγώ θα ήθελα να καταθέσω μια ερώτηση ως προς την κοινή γεωργική πολιτική. Έκανε κάποιες προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το πρασίνισμα. Μας είπατε ότι θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της Επιτροπής οι συζητήσεις. Όσον αφορά όμως τα ερωτήματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπιστώνουμε μεγάλη διαφορά απόψεων μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν κράτη τα οποία ιδιαίτερα φροντίζουν τους γεωργούς τους, τους κτηνοτρόφους τους, μετά από αλλού ακούγεται ότι θα αυξηθούν το κόστος. Ανακοινώνονται διάφορες πρωτοβουλίες, αλλά τίποτα συγκεκριμένο δεν βλέπουμε. Άρα θα πρέπει, πιστεύω, να γίνει τώρα μια προσπάθεια με ένα φόρουμ συζητήσεων μεταξύ γεωργών και κυβερνήσεων. Μια άλλη ερώτηση που ήθελα να διατυπώσω. Λόγω περιεργίας. Διαπιστώνουμε διαφορετικό επίπεδα ποιότητας σε τρόφιμα που κυκλοφορούν στις αγορές διαφορετικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι, είναι, ότι υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ποιότητας δεν ξέρω αν έχετε ακούσει εσείς τέτοιες συζητήσεις, αν έχετε παρακολουθήσει τις συζητήσεις και αν έχετε κάποια γνώμη γι' αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάντμπαχ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Επί της ουσίας η κυρία Υπουργό αναφέρθηκε σε ένα θέμα που με ενδιαφέρε πάρα πολύ ως προς την μικροβιακή αντίσταση. Αλλά δεν ήθελα να προχωρήσω λίγο περισσότερο, διότι πριν από μερικές ημέρες ε, ενημερωθήκαμε για μια μελέτη λάβαμε γνώση μιας μελέτης που λέει ότι από τη Σουηδία όπου γίνεται επεξεργασία διαφόρων υφασμάτων ε, με αντιμικροβιακό υλικό, κατά το πλήσιμο το υλικό αυτό περνάει μέσα από το πλυντήριο στα, ε, στην αποχέτευση και τους υδατινούς πόρους στη συνέχεια, στο περιβάλλον γενικότερα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω κύριε Υπουργέ, εάν έχετε κάτι συγκεκριμένο και εσείς αν έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό, φέρει δύο κτώνα. Έχετε, έχετε υπόψη να παρακολουθήσετε την υπόθεση αυτή πιο στενά. Γιατί ναι βεβαίω υπάρχει μια, ένας κανονισμός ο οποίος επιβάλλει την υποχρέωση για επισήμανση όταν ε, περιλαμβάνονται οκτώνα κάπου, αλλά δεν προβλέπεται τίποτα όσο προς την περίπτωση που αυτά περνούν στο περιβάλλον μέσω του πλησίματος. Και επίσης οι μικροίνες, γενικά τα μικροιλικά τα οποία μπορεί να μπαίνουν ακόμη και μέσα στην τροφική μας αλυσίδα. Ε, πώς σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάντμπαχ. Κύριο Σνέλχαρτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία σας εδώ ε, μας ε, κίνησε το ενδιαφέρον και ήταν πολύ φιλόδοξα τα όσα μας είπατε. Ωστόσο βλέποντας ε, τα θέματα που έχετε να αντιμετωπίσετε μπορούμε νομίζω να ανησυχούμε κάπως στην Ευρώπη γιατί εκ παραλλήλου και με τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική κρίση πολλά είναι τα ζητήματα τα οποία πιστεύω δεν ε, θα προχωρήσουν σε εφαρμογή όπως δεν έχουν μέχρι τώρα προχωρήσει σε εφαρμογή τα κράτη-μέλη και είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε πιστεύω διεξοδικά για την γεωργική μεταρρύθμιση Φερρυπίν, ένα παράδειγμα είναι η ε, διασταυρούμενη συμμόρφωση. Ε, δεν συζητάει όμω κανεί για άλλα ζητήματα, για ζητήματα ασφάλεια των τροφίμων κτλ. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώ σκοπεύετε να επιλύσετε τα προβλήματα αυτά, ενδεχομένω και συνεργασία με τον Επίτροπο των Αρμόδιων για την Ενέργεια και για την ε, Γεωργία. Η βασική αρχή τη αγρανάπαυση για το πρασίνισμα, η κάλυψη του κόστου ε, που έχει τόσο πολύ σημαντικά αυξηθεί τα τελευταία χρόνια για την αγρανάπαυση αυτή και το πρασίνισμα τη γεωργία. Πώ πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί, χωρί να θέλω βεβαίω να αμφισβητήσω την ιδέα του πρασινίσματο τη ε, γεωργία, των αντίον μάλιστα πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε και τα μέσα τα οικονομικά για να την εφαρμόσουμε. Αυτό λοιπόν δεν το συζητούμε. Συζητούμε πάντοτε προς μια κατεύθυνση αλλά δεν αναγνωρίζουμε ό,τι φαίνεται τα προβλήματα. Μεταφορές μεταφορές. Πολλές είναι οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα που έχουμε εγκρίνει εδώ στο Κοινοβούλιο. Και τώρα βλέπουμε ότι ακολουθείται μία γραμμή, γραμμή που εξετάζει μόνο το χρόνο μεταφοράς. Αλλά όποιος ασχολείται με την ε, ψυχολογία των ζώων γνωρίζει ασφαλώς ότι το σημαντικό κριτήριο δεν είναι το πόση ώρα ταξιδεύει ένα ζώο, δεν προξενεί αυτό το περισσότερο στρες, αλλά πόσες, ε, τι άλλες συνθήκες μεταφορών υπάρχουν, Φερρυπίν, τι είδους τι είδους φόρτωσης, εκφόρτωσης υπάρχει, με τι είδους όχημα μεταφέρεται. Επομένω δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε το ζήτημα της μεταφοράς των ζώων και της επιμαρίας των, των ζώων κατά τη μεταφορά στην ε, ποιότητα και μόνο του ε, στο, στη διάρκεια και μόνο της μεταφοράς πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία συνολικά. Διαφορετικά παραγνωρίζουμε το πρόβλημα. ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα σχέση με τα αντιβιωτικά και την ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πάνω απ' όλα στον ε, χώρο των νοσοκομείων, της νοσοκομιακής περίθαρψης. Εάν δούμε μια, ε, τη συνταγή που δίνει ο γιατρός για κάποιον που έχει ένα σχετικά ε, ισχνό οργανισμό, ένα σχετικά ισχνό σώμα και αντίστοιχα σε κάποιον άλλον πολύ πιο σωματώδη, δίνει το ίδιο δισκείο αντιβιωτικού. Είναι δυνατό να είναι αυτό ε, σωστή συνταγή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια προσαρμογή ως προς το, το βάρος, τη μάζα πάντων του ασθενούς. Κάτι άλλο που ενδιαφέρει ιδιαίτερος ε, τον πολίτη είναι ε, η ημερομηνία λήξεως των προϊόντων. Όταν βλέπει δηλαδή μια ημερομηνία τελευταία χρήση του προϊόντο ο καταναλωτή ε, ξέρει ότι πρέπει να το πετάξει και να μην το καταναλώσει. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα τη ασφάλεια των τροφίμων και νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ. Η κυρία Λίντα Μακέβαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, για όλα τα Ωραία που μας είπατε. Μας μιλήσατε για την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Το έχουμε συζητήσει και εδώ και ξέρετε υπήρξε μεγάλο λόμπι να μην μιλήσουμε για τα φάρμακα που παίρνουν τα ζώα. Ενώ πρόκειται για μια πραγματική ανησυχία που έχουν επαγγελματίε. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε και τις δύο αυτές πτυχές και την κατάχρηση που γίνεται ε, από τους ανθρώπους αλλά και από τα ζώα που πολλές φορές τους δίνουμε υπερβολικά πολλά αντιβιωτικά. Όντως, όπως είπαν και άλλοι και ο Chris Davids, όντως είναι πολύ σημαντικό το, το ένα εκατομμύριο υπογραφές που έχουμε μαζέψει και για την αλία όμως ισχύει το ίδιο. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε τους υπουργούς. Δεν είναι τεράστιο θέμα αυτό αφού ενδιαφέρει τόσο πολύ κόσμο. Πριν από λίγο καιρό μπορεί να μην φαινόταν ότι ε, ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι μόνο τους νοιάζουν τα λεφτά που πάνε, τους ενδιαφέρει. Και ούτε μπορούμε να κατηγορούμε πάντα τις Βρυξέλλες. Σαν να μην είχαμε πρόβλημα με την αλία νωρίτερα, με την μείωση δηλαδή των αποθεμάτων. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, ήδη από τη δεκαετία του 50 και του 60 είχαμε πρόβλημα μείωση των αποθεμάτων. Τέτοια πράγματα λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας ε, εν ώψη της μεταρρύθμισης. Τώρα, οι έλεγχοι που γίνονται στο κρέας. Ναι, υπάρχουν εδώ και άλλοι που είναι ειδικοί σε αυτό. Ξέρω ότι κατά το παρελθόν υπήρξαν κινήσεις που έγιναν ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν περισσότερο λόγο. Να έχουν δηλαδή και τους δικούς τους επιθεωρητές. Το έχουμε συζητήσει αυτό κατά το παρελθόν εδώ. Εμείς θέλουμε ανεξάρτητους ελεγκτές, ανεξάρτητους από τις επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι πραγματικά ανεξάρτητοι οι ελεγκτές οι οποίοι δουλεύουν για την επιχείρηση την οποία ελέγχουν, πόσο κάνεις να είναι πραγματικά ανεξάρτητοι. Τέτοιους θα έπρεπε όμως να χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο στο κρέας. Ευχαριστούμε, κύριε Μακάβεν. Επόμενος, η Γιούλη Γέλινγκ. Α, δεν τη βλέπω. Η κυρία Όκαν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, και εγώ θα μιλήσω δανέζικα μαζί σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Είναι μεγάλη χαρά να σε βλέπουμε εδώ και εννοείται ότι οι προσδοκίες μας είναι μεγάλες. Γι' αυτό και θέλω να αναφερθώ σε δύο πράγματα τα οποία συζητιούνται πολύ τελευταία. Το ένα είναι τα novel foods, τα νέα τρόφιμα. Το συζητάμε πολύ διότι η Κομισιόν, η Επιτροπή και μέρος του Συμβουλίου το έχει καταλήψει. Εγώ πιστεύω ότι εδώ πέρα υπάρχουν συμφέροντα του κλάδου που μπορεί να μην είναι καθαρά ευρωπαϊκά, αλλά διάβασα ένα άρθρο στη Herald Tribune και υπάρχει η Ισπανία, η Σουηδία που έχουν συμφέροντα εκεί. Η Δανία παίζει ιδιαίτερα επικοδομητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Η... Πρέπει να πούμε λοιπόν στην Επιτροπή ότι πρέπει να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θέλουμε επίσης απαγόρευση και όσον ε, αφορά τα ζώα αναπαραγωγής. Αν η νομοθεσία πρέπει να έχει κάποιο νόημα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους απόγονους, δεν ξέρω, μία, δύο γενιές. Δεν ξέρω πού πρέπει να σταματήσουμε. Για το θέμα της ανιχνευσιμότητας, η Επιτροπή μας είπε ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις, για να το πω έτσι. Να λοιπόν, τι πρέπει να προωθήσουμε. Υπάρχει και η νανοτεχνολογία. Ίσως και αυτό θα έπρεπε να μπει στην ημερήσια διάταξη της Δανέζικης Προεδρίας, γιατί είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει καλά. Θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί και ελπίζουμε ότι θα έχετε την ευκαιρία να ξεκινήσετε τη συζήτηση γι' αυτό. Κάτι άλλο τώρα. Δεν απαντήσατε στην ερώτηση του Κάρλ Σλούτερ για τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Και δεύτερον, κάτι που αφορά τη Δανία, που συζητάμε στην Επιτροπή Αναφορών, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα μύδια στα φιόρδ. Ξέρω ότι η Κομισιόν έχει απαντήσει σε αυτό. Ε, στη Δανία κάναμε κάτι το οποίο απαγορεύεται σε άλλες χώρες που έχει να κάνει με τις ζώνες του Natura 2000. Βέβαια αυτό στοιχίζει σε θέση απασχόλησης, μπορεί να είναι κρίμα, αλλά πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Δεν θα πρέπει να δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης σε βάρος των ε, τοποθεσιών του Natura 2000. Ξέρουμε ότι υπάρχει αλία σε ευάλωτα ύδατα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε την προστασία των υδάτων αυτών. Αλλά ιδιαίτερα το θέμα της κλωνοποίησης με ενδιαφέρει πόσες γενιές μετά δηλαδή προχωράμε και το θέμα αυτό της Δανίας. Ευχαριστώ. Φλόρενς και μετά ο Σλούτερ που έχει μια συμπληρωματική ερώτηση. Φλόρενς πρώτα. Ευχαριστώ πολύ και κυρία Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Πολλά είναι τα ερωτήματα που δεν μπορούμε να θέσουμε βέβαια όλα. Είχαμε μια διαδικασία συνδιαλλαγής με το Συμβούλιο. όπου είχαμε μια καταστροφή ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούσε κανείς να συνομιλήσει με κανέναν, δεν ασχολούνταν κανείς με την προσπάθεια για συνδιαλλαγή. Καθένα καθένας από τη δική του πλευρά και το μόνο που θα μπορούσα να πω ήταν να σας ανθαρρύνω, να δείξετε θάρρος, να αντιμετωπίσετε με παρησία αυτό το πράγμα και πάνω απ' όλα να κάνετε προτάσεις υπέρ της Ευρώπης της ίδιας. Δεν μπορεί κανένα κράτος να παραβλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση αλλαγή ούτε η δική μου η πατρίδα ούτε κανένα άλλο κράτο έδειξαν ε, βούληση να ε, στηρίξουν την ευρωπαϊκή προοπτική, να δώσουν ευρωπαϊκές λύσεις δηλαδή και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει η Προεδρία να διαδραματίσει τον δικό της ε, σημαντικό ρόλο. Δεύτερον, και με έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό, είναι το ζήτημα της αυξανόμενης συγκέντρωσης χώρων διάθεσης, πώλησης μεγάλων κέντρων ε, της κτηνοτροφικής παραγωγής. Οχτώ επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες στη Γερμανία αγοράζουν ε, το 80% της παραγωγής χοιρινού κρέατος, σε παραδείγματι. Άρα ελέγχουν ένα τεράστιο κομμάτι της αγοράς και προφανώς μπορούν και τους ε, κανόνες και τις διατάξεις να παραβλέπουν, να παραβιάζουν και υπό ε, καθεστώς συσκότησης να ε, δρούν όταν το επιθυμούν. Έχετε λοιπόν εσείς κάποιες συγκεκριμένες ε, προτάσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε Γιατί βέβαια αν δει κανεί ε, να πουλιέται στο ράφι του σούπερ μάρκετ ένα κοτόπουλο ε, στο, στην τιμή των 2 2 ε, ευρώ και 60 λεπτών. προφανώς κάτι δεν πάει καλά. προφανώς δεν τηρούνται κάποιοι κανόνες, Δεν θα πρέπει λοιπόν να παρεμβούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θα έπρεπε φερειπή να διεκδικούμε καλύτερη οργάνωση της διάθεσης στην αγορά, να παραμένει πιο μέσα σε πιο στενά τοπικά όρια, τοπική παραγωγή σε τοπική ε, διάθεση. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για την μεταφορά των ζώων των ζώων. Συμφωνώ μετά όσο είπε ο κύριο Νέλχαρτ, αλλά ω προ ε, το οχτάρο τη μεταφορά έχω διαφορετική ε, θέση, γιατί έχω και γεωργική δραστηριότητα ο ίδιο, όπου Βεβαίω πρέπει να πω ότι ε, οι συνθήκε μέσα στη Γερμανία είναι διαφορετικέ από ό,τι φερειπίνει τη Δανία. Γιατί αν η Δανία θέλει να πουλήσει, να ε, ζώα κρέα στην Ισπανία, δεν μπορεί να το πουλήσει με τη μορφή ζώντο ζώου και να τα μεταφέρει από την Δανία μέχρι την Ισπανία με φορτηγά, αλλά μάλλον σε μορφή σφαγίου μπορεί να το πουλήσει μόνο. Είναι λοιπόν ίσω διαφορετικέ λύσει που θα πρέπει να δίνονται ανάλογα με την περίπτωση. Και θα έλεγα ότι το, το δυστύχημα στην υπόθεση αυτή είναι ότι καθοδηγεί, ότι δίνει τις, ε, λαμβάνει τις επιλογές, δίνει τις, ε, επι, τις επιταγές της ή τις διαταγές της ίδια η βιομηχανία κρέατος και όχι ο καταναλωτής, όχι η πολιτεία. Αισθανόμαστε όλοι πολύ αδύναμοι όταν βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση στην αγορά, ειδικά εμείς, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου που είμαστε μέσα στην αγορά αυτή. Ευχαριστώ. Κύριε Σλίτερ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τις πιο δίκαιες τιμές και για τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, δεν είναι θέμα μόνο χρήσης της γης. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Στην ε, άτυπη συνάντηση 3 και 5 Ιουνίου, τι θα λέγατε να προσκαλέσετε όλους τους ευρωβουλευτές και όλους τους υπουργούς να μεταφερθούν ε, στην Κοπεχάγη κάτω από τις ίδιες συνθήκες <laughs> όπως μεταφέρονται και τα ζώτα ζώα. Να καλέσουμε όλους τους υπουργούς και όλους τους ευρωβουλευτές και εμείς με τις ίδιες συνθήκες όπως μετακινούνται τα ζώα έτσι να, μετακινου... μετακινηθούμε και εμείς και να δούμε πόσο πολύ θα μας αρέσει αυτό. Ωραία κύριε Σλούτερ. Ο κύριος Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Ξέχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα γιατί έχω και το θέμα της ε, ε, γενετικής τροποποίησης ως εισηγητής αναλάβει και θα ήθελα να ρωτήσω Μπορούμε να περιμένουμε μια συγκεκριμένη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή ή θα πρέπει να κάνουμε ε, μια άλλη κίνηση. Γιατί στο θέμα της υγειονομικής, ε, της υγιεινής των ζώων ε, δεν μπορούμε να ε, παραμελήσουμε πολλά από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Έχουμε ζήτημα φερρυπίν ως προς τα σφάγια, προς τη σφαγή των, ζώων, ως προς την παρουσία ζωονόσων ή άλλων, άλλης μορφής κινδύνων και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω πότε και τι πιστεύετε ότι μπορούμε να περιμένουμε και αν, αν θεωρείτε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε μέσα στη θητεία σας, δηλαδή μέσα στην προεδρία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και το δεύτερο κύριο ερωτήσεων. Η υπουργό έχει το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ για όλες τις καλές ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι δύο τις έχω ξεχάσει ίσως να μην... Ε, Τη σημείωσα την πρώτη φορά. Μη, ε, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Η απόφαση προς το παρόν για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς η πρόταση είναι στο Συμβούλιο όπου θα εξεταστεί το Μάρτιο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξη. Πάντως η Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί με τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την πρόταση αυτή των Βρυξελών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση, αλλά θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια συζήτηση και διαπραγματεύσεις. Εκεί βρίσκεται η Προεδρία όσον αφορά αυτό το θέμα. Για τα νέα τρόφιμα τώρα. Η Μαγκριτ Άλκεν ρώτησε για την κλωνοποίηση και για την ανεχνησιμότητα. Και εδώ περιμένουμε ότι περιμένουμε πρωτοβουλία από την Κομισιόν. Εκεί βρισκόμαστε. Κύριε Άκεν, όχι στη βία, ε. όχι με το ζόρι. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Τι να σας πω, περιμένουμε αυτή την πρωτοβουλία. Όσον αφορά τώρα τα μύδια στα δανέζικα φιόρδο, αν δεν έχετε αντίρρηση, ας το συζητήσουμε διμερός, διότι δεν έχω να κάνω σχόλια της Προεδρίας για αυτό το θέμα. Κυρία Μακάβεν, αναφέρεστε στα αντιβιωτικά και την κατάχρηση που γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να επικεντρωθούμε όταν πρόκειται για αυτό το θέμα και στην κτηνιατρική πτυχή αλλά και στην ανθρώπινη υγεία. Και τους δύο τομείς πρέπει να τους εξετάσουμε και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και στους δύο τομείς. Σημαντικό αυτό. Αναφερθήκατε και στην αλία, το ότι την χρειαζόμαστε θα γίνει συζήτηση στην υδατοκαλλιέργεια, στο Συμβούλιο Υδατοκαλλιέργειας θα συζητηθεί. Πώς να έχουμε δηλαδή βιώσιμη, ε, αηφόρο, εννοείται ότι έτσι πρέπει να είναι η υδατοκαλλιέργεια. Τώρα για τους ε, ιδιώτες ελεγκτές. Έτσι, αναφερθήκατε στον έλεγχο του κρέατος. Το βασικό για τον έλεγχο αυτό τον πρώτων κρέατος είναι να έχουμε μια ρύθμιση η οποία θα διασφαλίζει ότι η επιθεώρηση είναι αξιόπιστη, ότι ο έλεγχος είναι αξιόπιστος, ότι έχουμε τους ελέγχους που χρειαζόμαστε. Μερικές φορές, εντάξει δεν νομίζω ότι υπάρχουν συμπεράσματα του Συμβουλίου για το κατά πόσο ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Το βασικό είναι να γίνεται ο έλεγχος. Πάντως θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια τη Δανέζικη Προεδρία η αποτελεσματικότητα των ελχώνων αυτών. Τώρα, η, τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Κύριε Φλόρενς, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Είχαμε μια σχετική οδηγία, γίνανε πολλές συζητήσεις, συμφωνώ, αλλά από πλευράς επίσημα της Προεδρίας δεν μπορώ να σας πω κάτι. Προσωπικά μπορώ να σας πω ότι έχει τεράστια σημασία να μπορούμε να αποσύρουμε τα μέταλλα και τα συστατικά τέλο πάντων των ε, ηλεκτρικών συσκευών και αν μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε και να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Επιτρέψτε μου εδώ να σας μιλήσω όχι από την ιδιότητα της Προεδρίας, αλλά ως ε, πολιτικός που μιλάει σε άλλους πολιτικούς. Πολλοί από εσά ανηφέρθηκαν στα διλήμματα που έχουμε όσον αφορά τις χημικές ουσίες. Ε, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε πρόβλημα με τη χημεία, με τα χημικά. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι επηρεάζουν τη δυνατότητά μας να κάνουμε παιδιά. Και υποφέρουμε από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε στέρες επιστημονικές γνώσεις για αυτό το θέμα. Και Εκεί είναι που εγώ έχω ανησυχίες ως πολιτικός. Διότι φοβάμαι ότι σε 20 χρόνια ο κόσμος θα έρθει και θα μου πει «Ήσουν εκεί, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας και θα μπορούσες κάτι να έχεις κάνει». Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για τα χημικά να έχουμε τεκμηρίωση για να μπορούμε έτσι να σταματάμε οτιδήποτε είναι βλαβερό και επικίνδυνο για την υγεία μας που μειώνει τις δυνατότητες ε, ε, των ανθρώπων να κάνουν παιδιά. Τώρα, το επίσημο που έχω να πω είναι ότι έχουμε μια πριγκίπισσα στη Δανία και φυσικά θα θέλει να κάνει παιδιά. Χαίρομαι. Σήμερα το πρωί μάθαμε τα νέα, φαίνεται ότι ετοιμάζεται. Τα πράγματα προχωρούν, βλέπετε, σε ορισμένες υποθέσεις, τουλάχιστον στην βασιλική οικογένεια της Δανίας. Επίσης αναφερθήκατε στο πρασίνισμα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Φυσικά, ποια είναι τα δύο στοιχεία εδώ. Το ένα είναι να έχουμε πραγματικό πρασίνισμα και το άλλο είναι να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας για την ΚΑΠ. Δεν ξέρω τι γίνεται σε εσά. Έχουμε 45.000 που παίρνουν επιδοτήσεις στη Δανία και αν πρέπει να τους υποβάλω σε 170 ερωτήσεις για να πάρουν τα χρήματά τους, ε, αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον οι ορθές. Να έχουμε ρύθμιση και έλεγχο, αλλά και λιγότερη γραφειοκρατία όσο γίνεται. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ, για τα πολύ σαφή λόγια που μας απευθύνατε για τις ε, πολύ σαφείς δεσμεύσεις και για τη θεματολογία βεβαίως ε, που τόσο πολύ ενδιαφέρει τον πολίτη όπως οι μεταφορές των ζώων ε, θα έχετε εσείς κατά την θητεία σας την ευθύνη αυτή και να ανταποκριθείτε δηλαδή σε μια πρωτοβουλία πολιτών. Και δεν είναι μόνο αυτή, ε, εμείς ως Κοινοβούλιο θα έχουμε την ευκαιρία να ε, κάνουμε μια ακρόαση στην οποία και η Επιτροπή αλλά βέβαια και το Συμβούλιο θα είναι προσκεκλημένη και πιστεύω ότι θα ελπίζω ότι θα έχουμε στο δυνατόν καλύτερη εκπροσώπηση από τη δική σας ε, Προεδρία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Να ε, είσαστε βέβαια για τη δική μας την υποστήριξη. Θα είμαστε στο πλευρό σας ε, στην πορεία αυτή, στο Συμβούλιο, για να έχουμε σωστές επιλογές και όχι μόνο γραφειοκρατικές, αλλά και πάνω απ' όλα για να έχουμε αποτελέσματα βιώσιμα και διαρκή δεν ξέρω πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε ως προς την επιτυχή διαξαγωγή των εργασιών του, ε, του Συμβουλίου, αλλά πάντως είμαστε στο πλευρό σας ε, ε, στην πορεία αυτή. Εάν χρειάζεστε οτιδήποτε, είμαστε στη διαθέσή σας. Και ξέρω ότι θα είναι μια κουραστική ε, περίοδος, αυτό εξάμεινο, αλλά πάντως είμαι βέβαιος ότι θα στεφθεί και με επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you So, die Sitzung ist dann unterbrochen. Wir fangen pünktlich um 15 Uhr wieder an mit einem. Τελειώνει η συνεδρία τώρα, μάλλον διακόπτεται εδώ. Ξαναρχόμαστε ακριβώ στι 3 και παρακαλώ του συναδέλφου να στην ώρα του έχουμε πάλι υπουργό.